So, Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Σήμερα έχουμε διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν είναι η Ένωση Καινοτομίας, η Ευρώπη μετά την κρίση. Η κυρία Μέρκης είναι η συγγήτρια, υπάρχουν και διάφοροι σχιώδεις συγγητές και η κυρία Μέρκης ξεκινάει καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρόκειται για το θέμα το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσει την, ε, τις προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, και ιδίως την έλλειψη ενεργείας για να έχουμε μία νέα κατάσταση. Βεβαίως πρέπει να ε, να ασχοληθούμε με τα βασικά θέματα και να προσπαθήσουμε ε, να λύσουμε το πρόβλημα της κρίσεως. Βεβαίως, συνήθως μιλάμε ε, για ένα τρίγωνο για τις κυβερνήσεις και δεν ε, θέλω να αναφερθώ σε άλλα θέματα αλλά ε, αυτό που θεωρώ είναι ότι η πιο βασική καινοτομία δεν έχει ε, ε, ληφθεί υπόψη και στο κάτω-κάτω, εάν ε, οι ε, πολίτες δεν μας ακολουθήσουν στην προσπάθεια καινοτομία δεν θα υπάρξει καινοτομία, οπότε πρέπει να ασχοληθούμε καταρχήν με τις ε, απαιτήσει των πολιτών. Άρα είναι η εξουσία των πολιτών. Αυτό είναι το βασικό θέμα της ενώσεως της καινοτομίας μας. Επίσης, ήδη ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα νέο μέσο την, ε, την εταιρική σχέση με τους ε, με τους πολίτες και την ε, συνεργασία κατά τρόπον ώστε να υπάρξει ε, ανταπόκριση. Ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Είχαμε μία πρώτη μια πρώτη ε, συζήτηση επ' αυτού, μια πρώτη επικοδομητική συνεδρίαση και ήταν σαφές ότι ε, πρέπει να υπάρξει τυποποίηση και χρηματοδότηση και αυτά είναι τα πιο βασικά θέματά μας. I there is no label on social innovation. So what I would very... Αυτό λοιπόν που θα ήθελα ε, είναι να μην ασχοληθούμε μόνο με την γενική ε, θεωρητική ε, αντιμετώπιση αλλά να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα ε, βήματα για να μπορέσουμε να υποκινήσουμε την καινοτομία. Η καινοτομία είναι σημαντική. Είναι όμως πολύ σημαντικό στην Ένωση της Καινοτομίας να καθορίσουμε τι σημαίνει ακριβώς καινοτομία. Διότι υπάρχει πάντοτε δυνατότητα να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, αλλά περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για μία διαδικασία πρόκειται για τρόπους με τους οποίους θα αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας γιατί νομίζω ότι έχουμε ε, θεωρήσει ότι πρόκειται ε, για ε, ένα προϊόν μίας διαδικασίας ερευνητικής. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μπορεί να αλλάξει τα διάφορα, ε, ε, τις διάφορες δυνατότητες ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να τροποποιήσουμε και την κοινωνία δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα και πολλοί των οποίων η ουσιαστική εργασία είναι η ενέργεια και θα πρέπει να ε, δώσουμε πιο μεγάλες δυνατότητες και ενοτομίες στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή ζωή των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η ε, Ένωση της Καινοτομίας ε, έχει στενή συνεργασία ε, με το, την αυαρχίδα της βιομηχανικής πολιτικής όπου η ψηφιακή, το ψηφιακό πρόγραμμα και, ε, το, ε, και η ναυαρχίδα της αποτελεσματικότητας συνδέονται στενά. Θέλω λίγο να σχολιάσω την ενιαία αγορά, διότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και μας ανησυχεί περισσότερο είναι η ενιαία αγορά. Έχω δει τόσα πολλά παραδείγματα καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων που δεν μπορούσαν να, να ε, εξάγουν τα προϊόντα του τους λόγω διαφορετικών συστημάτων και διαφορετικής φορολογίας και διαφορετικών υγειονομικών διατάξεων που δεν επέτρεπαν να, τα καινοτόμα αυτά προϊόντα να εισαχθούν σε μια νέα αγορά. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να συνδυαστεί ε, η καινοτόμος αγορά με την ε, ε, ε, Ένωση την και να την ανανεώσει και να, την, ε, να υπάρξει μία καινοτομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε αυτό το οποίο ε, εγώ ζητώ στηρίζεται και από πολλούς συναδέλφους. Χρειαζόμαστε δηλαδή μία πιο ενιαία πολιτική ε, και ένα συντονισμό με τις διάφορες άλλες πολιτικές για να δούμε πώς θα προωθήσουμε την ενιαία αγορά και πώς θα προωθήσουμε την καινοτομία. Βέβαια και η κυβέρνηση είναι ένα σημαντικός παράγον. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δημόσιες αγορές, διότι οι δημόσιες αγορές είναι πολύ σημαντικές για να προωθήσουν την καινοτομία και ε, ένα καλό σύστημα για ευρωπαϊκές ε, για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για να υποκινήσουμε ε, την αγορά είναι ε, να ε, συνδυάσουμε αυτές τις προσπάθειες με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία. Πώς θα προωθηθεί και η καινοτομία. Είχαμε πει στο παρελθόν ότι 3% του ΑΕΠ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για έρευνα, έρευνα και ανάπτυξη και ο Επίτροπος ήδη μας είπε ότι θέλει να μετρήσει ε, την, ε, τη διεργασία μέσω των αποτελεσμάτων. Τι είναι όμως τα αποτελέσματα, πόσο θα ε, μετρήσουμε την καινοτομία, πρέπει να καταρτήσουμε ένα κατάλογο δικτών. Θα ήθελα λοιπόν πριν τελειώσω να αναφερθώ στο ρόλο των περιφερειών στο πλαίσιο αυτό διότι οι περιφέρειες ε, μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία είναι πιο κοντά στις επιχειρήσεις και συνήθως και στις ε, ερευνητικές ε, εγκαταστάσεις οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις προωθήσουμε και βεβαίως δεν είχα απόλυτο δίκιο διότι είπα ότι θα ξεκινούσα από τις συνεργασίες αλλά πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε την καινοτομία και ε, πιστεύω ότι σε αυτό χωρίς να υπερβάλλω Πιστεύω ότι έχουμε 10 έως 20 ταμεία. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τις περιφέρειες να χτυπήσουν τη σωστή πόρτα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει συγχρόνως αυτό να απλοποιηθεί. Η απλοποίηση είναι πολύ σημαντική. Άρα αυτό το οποίο είπα όταν χρειαζόμαστε ένα one-stop shop τι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουμε ένα, ένα επίπεδο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν σε ποιο ταμείο πρέπει να απευθυνθούν και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χτυπώντας την πόρτα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα τους κατευθύνουν στο σωστό ταμείο. Θα μπορούσαμε ίσως να τους συνδυάσουμε με τους σωστούς συνεταίρους που επεξεργάζονται το ίδιο θέμα. Δεν μιλάω λοιπόν για ύπαρξη ενός μοναδικού ταμείου αλλά για μια υπηρεσία η οποία οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την κατάσταση χωρίς να έχει σημασία από πού έρχεται ο χρήστης υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι επεξεργάζονται αυτό το θέμα, ζητούν μία αναθεώρηση του συστήματος ε, χρηματοδότησης, να μην υπάρχουν πλέον επιδοτήσεις, αλλά ένα σύστημα αμοιβών, μπόνους και να υπάρξει συγχρόνως και ένας ε, τρόπος για να δούμε πώς ε, θα υποκινήσουμε την καινοτομία. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να συνεργαστείτε μαζί, του, μαζί μου για να δούμε πώς αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και τέλος όσον αφορά τις καινοτόμες συνεργασίας είναι νέο ή παλαιό εργαλείο. Ζήτησα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο να σχολιάσει ε, τις ε, καινοτόμες ε, συνεργασίες και της είπα μήπως ε, όπως λέμε στην Ολλανδία πρόκειται ε, ε, για παλιά παπούτσια σε μία μάλλον σε, για παλιό κρασί σε μία νέα σακούλα είναι κάτι πραγματικά καινούριο μήπως είναι μόνο ένα νέο όνομα είναι όντως πιο συνετό εταιρικό υπάρχουν επιπρόσθετες προσπάθειες. Δεν ξέρω ποια είναι η μορφή διακυβέρνησης γιατί αυτό το σύστημα θα λειτουργήσει καλύτερα. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και ε, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει για τις καινοτόμες συνεργασίες και ε, για το πόσο θα μπορέσει η Επιτροπή να εξετάσει πώς θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Ε, συγχρόνως έχουμε ήδη τη συνεργασία για την ε, ε, υγιή γύρανση. Έχουμε πολλά, πολλές συνεργασίες καινοτόμες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ολόκληρο τον κατάλογο. Υπάρχουν όμως και πιλωτικές δράσεις και πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των πιλωτικών δράσεων. Αλλά αν υπάρξει ένας μακρύς κατάλογος αυτών των συνεργασιών θα υπάρχει κατακαιρματισμός και αυτό το οποίο ουσιαστικά εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι αλλαγές της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι θα υπάρξουν διάφορα θέματα που είναι πολύ ε, χρήσιμα ε, για όλους μας και ελπίζω θα μας δώσουν και νέες ιδέες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή στο θέμα και ο πρώτος που ζήτησε το λόγο είναι ο κύριος Τουσνόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σχολιάσω ε, τα όσα είπε η συγγήτρια, γιατί ως κοιόδης θεωρώ πως η συζήτηση που κάνουμε είναι πραγματικά ζωτική σημασία. Η καινοτομία αναμφίβολα είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για να προωθήσουμε και να επιταχύνουμε όλη τη διαδικασία ανταγωνιστικότητας τις βιομηχανίες μας. Γιατί βέβαια στον κύκλο της καινοτομία έχουμε μείνει πίσω και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο για να εισάγουμε την καινοτομία στην ε, παραγωγική διαδικασία από ό,τι στι Ηνωμένε Πολιτείε ή σε άλλου χώρου ανταγωνιστέ. Πρέπει να σα πω πω ε, η καινοτομία πρέπει να εισαχθεί σε όλου του χώρου στου οποίου ανέφερε η συγγήτρια και πιστεύω πω αυτή η πολύ γενική και διευρυμένη προσέγγιση είναι η σωστή. Ε, έχω βέβαια κάποια σχόλια πιο συγκεκριμένα. Ε, δημόσιες συμβάσεις. Δημόσιες προμήθειες, με συγχωρείτε. Το είπε άλλωστε και η συγγήτρια. Ε, νομίζω ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την στήριξη της ανάπτυξης. Αυτό βρίσκεται και στην έκθεση που έχουμε υποβάλει εμείς και Ακούστηκε και μια ρητορική ερώτηση για τα κατά πόσο θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτοκαθολικά. Ε, νομίζω πως ε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Φοβάμαι πως αν ορίσουμε τέτοιου αυστηρούς κανόνες θα οδηγηθούμε σε περιορισμό ε, των ενδεχόμενων αποτελεσμάτων γιατί ίσως αυτοί οι στόχοι να αποτελέσουν εμπόδιο ε, για τις ε, καινοτόμες προσπάθειες που θα κάνουν κάποιες περιφέρειες, κάποια κράτη, γιατί βέβαια αν θέσουμε ποσοτικούς στόχους θα δουν, α, πρέπει να συμμορφωθούμε, πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες με αποτέλεσμα να περιορίσουν το πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δράσεων που θα μπορούσε να καλυφθεί από τον όρο ε, καινοτομία. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν δεν θα βοηθήσουμε να επιταχυνθεί η έρευνα, και ούτε θα βοηθήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφερθούν στην ε, βιομηχανική παραγωγή. Στο δεύτερο σχόλιο για μια συζήτηση η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και για ένα κείμενο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω και εδώ το έχει σχολιάσει η ίδια η συγγήτρια, είναι η χρηματοδοτική διάσταση της κοινοτομίας. Δηλαδή, χρειάζεται να συζητήσουμε όλες ε, τις παραμέτρους τους θέματος αυτού. Δηλαδή πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία χρηματοδότησης της καινοτομία. Αυτό είναι και το πιο επίκαιρο θέμα και αυτό συχνά συνδέεται με την ανάπτυξη και την έρευνα και την ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας παραπέμψω πάλι στο τι κάνουν οι ΙΠΑ. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα σύστημα ταμείων μέσω του οποίου χρηματοδοτούμε, αλλά είναι προφανές πως αυτό το σύστημα ταμείων δεν έχει την απαραίτητη ευελιξία και μάλιστα τουλάχιστον σε επίπεδο γραφειοκρατία, είναι αρκετά δυσκίνητο. Θα έπρεπε λοιπόν να εξετάσουμε και κάποιε ακόμα δυνατότητε, ίσω έκδοση ομολόγων ή κάτι διαφορετικό, για να στηρίξουμε τι ερευνητικέ προσπάθειες, είτε αυτέ γίνονται στον χώρο τη τεχνολογία, είτε γίνονται στι κοινωνικέ επιστήμες. Νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως αποτελούν επενδύσεις υψηλού κινδύνου, γιατί κατά τη γνώμη μου το να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι θα μας βοηθήσει στο να, κάνουμε, ε, να παρουσιάσουμε περισσότερες καινοτομίες. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της καινοτόμου έρευνας να μεταφερθούν στην ε, καθημερινότητά μας είναι ένα διαφορετικό θέμα. Εκεί εμείς θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε όλο και περισσότερη γνώση να μεταφέρεται στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν ως σκιώδης ε, εισηγητής καλωσορίζω αυτή τη συζήτηση, θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά παράλληλα πιστεύω πως δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συζήτηση καθαρά φιλοσοφικού περιεχομένου, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς τα λεγόμενά μας μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια τα οποία πολλές φορές ε, παρεμποδίζουν ε, την καινοτομία στην Ευρώπη και επιμεκίνουν το χρόνο μετάφρασης της καινοτομίας σε αυτά πρακτικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να σας πω πως καταρχήν ευχαριστώ και συγχαίρω την κυρία Μέρκης γιατί οι προτάσεις της είναι εξαιρετικά φιλόδοξες για ένα θέμα το οποίο αποτελεί σημείο κλειδί για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αληθεύει πως η Ένωση για την Καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά, στον πυρήνα της ατζέντα για το 2020 και αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη και θα οριοθετήσει και τα όσα θα κάνουμε στο μέλλον. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε. Εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού προετοιμάσαμε μια γνωμοδότηση πολύ γρήγορα αλλά το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι μέσω της εκπαίδευσης, της παιδείας, της επιμόρφωσης θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σχόλια στο θέμα αυτό. Και πρέπει να σας πω πως εμείς έχουμε σχολιάσει και κάποια θέματα τα οποία πιστεύουμε πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και συζητώντας με την κυρία Μέρκης, νομίζω πως θα τύχουν καλής υποδοχής. Τρία σημεία λοιπόν είναι τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Η καινοτομία θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Δηλαδή, όχι μόνο τεχνολογική καινοτομία ή παραγωγική καινοτομία, αλλά που θα καλύπτει όλον τον οικονομικό χώρο και θα πρέπει η καινοτομία να ξεκινάει από, την, το αρχικό σπέρμα της ιδέας μέχρι το τελικό προϊόν. Δηλαδή η καινοτομία συνδυάζεται και συνοδεύει τη γνώση. Συνοδεύεται και από τη γνώση. Έχουμε πιο ανοιχτά, πιο ευέλικτα μοντέλα συνεργασίας, για παράδειγμα στις, ε, στην πολιτιστική βιομηχανία, που έχει ένα τεράστιο δυναμικό που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Θα πρέπει να στοιχηματίσουμε υπέρ ένα χώρο ευρωπαϊκό ε, πανεπιστημίων αριστείας στα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατόν επενδύσεις έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη συνέργεια μεταξύ των πανεπιστημίων και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερος βέβαια συνδυασμός και συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών κύκλων και ε, ακαδημαϊκών κύκλων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσει στέκονται πιο κοντά στον πολίτη και ε, στι επιχειρήσει. Θα πρέπει να σταθούν το ίδιο κοντά και στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε πω χωρί εκπαίδευση, χωρί άριστη μόρφωση, δεν έχουμε του πόρου που θα μα επιτρέψουν να επιτύχουμε του στόχου του οποίου θέσαμε στην ατζέντα τη Ευρώπη του 2020. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα είπε η κυρία Μέρκης σχετικά με τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες θα πρέπει να αποτελέσουν τον κοινό παρανομαστή όλων αυτών των ε, προσπαθειών. Αλλά για να είμαστε επιτυχημένοι εδώ θα πρέπει να σεβαστούμε ε, την λέξη εμπιστοσύνη. Η πλειοψηφία των πολιτών είναι κάπως διαφορετικά τα θέματα στη βιομηχανία, αλλά οι πολίτες δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει καινοτομία, δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους αυτούς και τους φαίνεται σαν κάτι μακρινό, σε μεγάλη απόσταση από τους ίδιους και θα πρέπει να τους εξηγήσουμε στην καθημερινή τους ζωή πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις καινοτομίε. Θα πρέπει να πιστέψουν στην καινοτομία και να αποκτήσουν περισσότερη γνώση. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη γνώση η οποία θα συνοδεύει ολόκληρη τη διαδικασία. Κάτι που είπε η κυρία Μέρκης είναι επίσης σημαντικό. Κοινωνική καινοτομία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να εντάξουμε εδώ. Αλλά εγώ θα τολμούσα να θέσω στο τραπέζι κάποια σημεία που έχουν να κάνουν με την κοινωνική καινοτομία. Για παράδειγμα, εξάλληψη της φτώχειας, βελτίωση της παιδείας και της μόρφωσης, ε, η μάχη κατά της εγκατάλειψης της, ε, ε, της σχολικής εκπαίδευσης και η πρόθεση του πολιτισμού. Ξέρετε πως η γνωμοδότησή μας από την Επιτροπή Πολιτισμού σύντομα θα φτάσει στα χέρια σας και όλες αυτές οι παρατηρήσεις σίγουρα θα ληφθούν υπόψη από την εισηγήτρια. Τσατσιμακάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία ήδη είχε συναντηθεί με τους σιώδης εισηγητές και έχουμε συνεργαστεί πολύ ε, στενά. Με ε, εντυπωσίαση ότι η Επίτροπος ε, Μακουίν έχει θέσει τόσο υψηλά στις προτεραιότητές της την καινοτομία και ε, μέχρι στιγμής ε, η έρευνα και η καινοτομία χωριζόντουσαν διατεχνητών μέσων και πρέπει να ε, διευκρινίσουμε ότι πρέπει να συνδυαστούν. Είναι και απαραίτητο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των ιδεών τους σε συγκεκριμένα προϊόντα ε, βρίσκονται σε υποδέστερη θέση από την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά η καινοτομία πρέπει άμεσα να ενταχθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για ένα επιπρόσθετο στοιχείο όπως ε, θεωρούν ορισμένοι διότι υπάρχουν πολλές ε, πολλές πτυχές ε, του χώρου της έρευνας αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό της έρευνας να είναι καινοτόμα διότι αν δούμε το τέταρτο ερευνητικό πρόγραμμα το 40% των προγραμμάτων γινόντουσαν με 40 με 40% ε, ε, συμμετοχή ε, των, της βιομηχανίας ενώ τώρα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ και βλέπω ότι η έκθεση της συναδέλφου αναφέρει τρεις φορές τη βιομηχανία και εννιά φορές τον κοινοτικό τομέα. Πρέπει να ξέρουμε για το τι μιλάμε. Μπορούμε να, ε, ε, να ε, χρηματοδοτήσουμε θαυμάσιες χαιρετόμες ιδέες αλλά πρέπει να αναλάβει κανείς και ορισμένους ε, κινδύνους να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε ε, ένα ποσοστό κινδύνου ε, διότι αν λάβουμε υπόψη το Skype το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με μέσω του ΤΣΙΠ και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ε, καταλήξαμε στο Skype το οποίο τώρα έχει ε, δημιουργήσει σε ένα είδος επανάσταση στον κόσμο. Λοιπόν, ε, στην ιδέα που έχουμε εδώ για την ε, Research Finance Facility RSFF ε, η Έρικα Μάν, που ήταν κάποτε συνάδελφός μας είναι η ομόλογό μας για το θέμα αυτό τώρα και υπάρχει πάρα πολλή καινοτομία για την οποία νομίζουμε ότι μπορούν να πλησιάσουν την αγορά να την επηρεάσουν αλλά θα πρέπει να τη συνδυάσουμε με ένα σύστημα όπως είπατε μπόνους ε, ανταμοιβή. Δηλαδή όταν κάποιος προκαλεί μια καινοτομία θα έχει το μπόνους αυτό διότι θα πρέπει να παίρνει το μπόνους αυτού μόνο όποιος όντως καινοτομεί και έτσι ε, θα αλλάξουμε την κατάσταση πρέπει όμως να αράρουμε ένα στοιχείο που ισχύει τώρα ε, όσον αφορά τη ο συνδυασμό με τη αδάνεια. Δηλαδή, εάν δεν κερδίσω μέσω της καινοτομία μου, δεν πρόκειται να αντιληφθώ και όλες τις δυνατότητες. Πρέπει να αποκλείσουμε την απαγόρευση κέρδους. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κέρδος. Και αυτό σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι πρέπει να διευρύνουμε τον ορισμό τον οποίο ήδη έχουμε καταρτήσει. Ε, διότι ε, βλέπουμε ότι ήδη έχουμε πετύχει ορισμένη μονοτομία, έχουμε αναστρέψει την κατάσταση, αλλά να ε, επικεντρωθούμε επιπλέον σε μεγάλα θέματα, ακόμη και για τις δημόσιες προμήθειες, που είναι θέμα το οποίο μας απασχολεί πώς θα διαμορφωθούν οι δημόσιες προμήθειες όπως στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή να υπάρχει ένα ποσοστό καινοτομία σε αυτό το τομέα. Δηλαδή αν, αν πούμε ότι στις δημόσιες προμήθειες χρειάζεται καινοτομία δεν θα ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε. Ενώ αν πούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 30% των μέσων για την τεχνολογία αποθήκευση στοιχείων ε, στους τομείς δηλαδή όπου ε, ε, Είμαστε πίσω από τους Κινέζους και από άλλους. Ε, αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε, να τους περιλάβουμε εις ε, τις ε, δημόσιες προμήθειες, να ζητήσουμε αύξηση της υψηλής τεχνολογίας και να επικεντρωθούμε σε δύο-τρία θέματα. Ο συνάδελφος Λάνιε, ευχαριστώ για να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα νομίζω ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα πλαίσιο δεν είναι ένας ε, δείκτης ότι πάμε καλά γιατί η βιομηχανία ε, έχει μεγαλύτερες ε, οικονομικές δυνατότητες από ό,τι εμείς με το πρόγραμμα πλαίσιο. Οπότε δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να καταρτήσουμε στρατηγικούς στόχους για την βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρώπη, να δούμε πού υπάρχουν ε, οι σωστές αγορές, πού υπάρχει το πλαίσιο που, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε και ποια πρέπει να είναι τα σημεία στα οποία θα ρίξουμε βάρος. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε ε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, δηλαδή στα στρατηγικά βασικά θέματα. Επιπλέον πρέπει να δούμε Πού χρειάζεται ουσιαστικά καινοτομία. Δηλαδή πέραν των ηγετικών προγραμμάτων της Ευρώπης πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τις περιφερειακές σχέσεις και τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου ε, οι μεγάλη, τα μεγάλα προγράμματα ε, δεν συμβάλλουν στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο όμως μπορεί να υπάρξει καλύτερη συνεργασία και γι' αυτό πρέπει να συνδυάσουμε την ε, διαρθρωτική πολιτική με την καινοτόμα πολιτική διότι ε, ε, υπάρχουν αποφάσεις πολιτικές ε, για επενδύσεις που εξαρτώνται από την καινοτόμα πολιτική. Οπότε ε, πρέπει να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις αυτές. Στην ε, κάτω Σαξονία αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμε ένα πρόγραμμα 60 εκατομμυρίων για καινοτόμες εφαρμογές και συμμετέχουν και τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις και ε, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με, τέτοια, με τέτοιους συνδυασμούς καλύτερα διότι δεν πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ε, ε, μόνο ότι η επιχείρηση ή ο ερευνητής πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμης της καινοτομίας αλλά και οι απασχολούμενοι δηλαδή θα πρέπει να βρούμε με τρόπο για να δούμε ε, πόσο θα ε, υπάρξει ε, η δυνατότητα να περιλάβουμε και τις δυνατότητες καινοτομία στα προγράμματα, πόσο θα εμποδίσουμε να υπάρξει μια άφηση των, της παραγωγής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η καινοτομία. Ευχαριστώ κύριος Λάμπερς. Ευχαριστώ. Πολλά έχουν υποθεί ήδη. Έχω καλυφθεί σε κάποιο βαθμό. Ε, ειδικά ταυτίζομαι με την παρέμβαση του κυρίου Χατζημαρκάκη. Για μένα η καινοτομία είναι ένα σύστημα όπου ε, πρέπει να διανοίξουμε τα σημεία συμφόρησης, να πιέσουμε, να λάβουμε ιδέες κτλ. Ξέρουμε ότι το επενδυτικό κεφάλαιο κινδύνου ε, στην Ευρώπη δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Ε, χρειάζονται και περισσότερες δημόσιες πρωτοβουλίες βέβαια, αλλά θα πρέπει να διευκολύνουμε και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να συνδυαστούν αυτά. Ε, και επίσης και να συνδυαστούν και με την περιφερειακή πολιτική, οι πολιτικές, ούτως ώστε ε, αυτά που κάνουμε σε επίπεδο ρυθμίσεων μέσω του επενδυτικού ταμείου να λειτουργήσουν και να επιταχυνθεί η συγκέντρωση επενδυτικού κεφαλαίου. Εάν δεν κινηθούμε στην Ευρώπη θα χάσουμε το τρένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, αν κινηθούμε δεν είναι σίγουρο θα τη στάσουμε, αλλά τουλάχιστον προ τα εκεί πρέπει, να κινηθούμε. Υπάρχουν πολλά σημεία συμφόρηση. επίσης. Στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών το αναφέραμε. Το θέμα των προτύπων. Η θέσπιση προτύπων είναι σημαντική. Ε, και μπορεί να σταματήσουν, αν θέτουμε, αν θέτουμε συνέχεια πρότυπα, μπορεί να σταματήσουμε την καινοτομία. Ε, Παραδείγματο χάρη, για την ηλεκτροκινητικότητα. Ε, αν δεν θέσουμε εμεί τα πρότυπα πρώτοι, θα τα θέσουν οι υπόλοιποι. Θα ήθελα λοιπόν γρήγορα, ταχαίω να θέτουμε τα πρότυπα. Εδώ ισχύει ο κανόνας 80-20. Εάν θέλεις να πετύχεις το τέλειο, το 100% ε, θα χρειαστούν αιώνε. Θα το κάνουν κάποιοι άλλοι αυτό που θα θέλει να κάνει εσύ. Πρέπει να συμβιβαστούμε γιατί και ο χρόνο είναι σημαντικό. Τώρα, το, καινο, το μοντέλο καινοτομίας στην Ευρώπη βασίζεται σε θέσπιση στόχων, ε, σε κανονισμούς, ε, σε πρότυπα. Έτσι ενθαρρύνουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Εδώ θέλω να ε, συνδέσω αυτά που λέμε τη συζήτηση που κάνουμε για, τις, ε, για την καινοτομία και τα αποτελέσματα που περιμένουμε από την καινοτομία. Το θέμα είναι να μην ε, πνίξουμε την καινοτομία με σωρούς, σωρία γραφειοκρατίας. Θα πρέπει απλώς εμείς να κινηθούμε και να απαντήσουμε στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις. Μίλησαμε για την καινοτομία. Ε, θέλουμε, βεβαίως το θέμα το, ένα άλλο θέμα είναι των πόρων, το θέμα της, ε, των δημογραφικών τάσεων. Ε, εδώ μπορούμε να μετρήσουμε, να βάλουμε στόχους ποσοτικούς. Εμείς ως ε, Επιτροπή Βιομηχανίας, συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουμε πιο αποφασιστικό και ηγετικό ρόλο. Όταν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, έχω στο μυαλό μου ακόμα και τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η Επιτροπή μας, η Ήτρε, ε, έχει μια δειλή και αμυντική στάση. Λέμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην είμαστε πολύ φιλόδοξοι, γιατί ο υπόλοιπος ε, κόσμος δεν κινείται τόσο γρήγορα και είναι σαν να αυτοτιμωρούμεθα. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά αν έχουμε χαμηλέ φιλοδοξίε, θα κάνουμε λίγα πράγματα. Οι υπόλοιποι δεν είναι κατά ανάγκη λίγο, λιγότερο φιλόδοξοι. Ορισμένοι είναι αρκετά φιλόδοξοι μάλιστα. Ακόμη και αν δεν θεωρήσουν ε, τους στόχους ε, δεσμευτικούς, θερυπίνοι οι Κινέζοι, όταν βάζουν στόχους, ε, οι Κινέζοι, οι υπόλοιποι, ο λαός ξέρει ότι πρέπει να τους σεβαστεί οπωσδήποτε. Δεν είναι ότι μου αρέσει το μοντέλο τους. Αυτό που λέω είναι ότι αν το παίξουμε πολύ αμυντικά, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε πρώτοι στο νήμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δείξουμε ηγετικέ τάσει. Δεν είναι η ώρα να κατεβάσουμε τα χέρια στο ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Το θέμα δεν είναι να υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε, είναι να κατακτήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ηγετικέ θέσει. Γι' αυτό, σε αυτό το επίπεδο, με αυτή την έννοια θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Μερικές φορές ε, πραγματικά μας δίνει την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα, αυτός εδώ είναι ένας χώρος που προωθούμε τις αμυντικέ α πούμε τάσει και λογικέ. Να το αναγνωρίσουμε συνάδελφοι ότι έτσι το παίζουμε. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες καλό θα ήταν να είναι πιο α, τολμηρές, πιο αφιλόδοξες, να παίρνουμε περισσότερους, περισσότερα ρίσκα. Ε, δεν μιλάω τώρα για λεπτομέρειες και για ανθυπο για ανθιπολεπτομέρειε. Για τα μεγάλα θέματα, α πούμε, για τι μεγάλε κοινωνικέ προκλήσει, εκεί πρέπει να είμαστε τολμηροί και φιλόδεξοι. Τώρα, για τι δημόσιε προμήθειε. Αυτό είναι ένα εργαλείο πολύ ε, σημαντικό. Το 17% του ΑΕΠ είναι δημόσιε ε, προμήθειες. προμήθειε. Σωστό είναι αυτό. Αλλά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και κριτήρια καινοτομία. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που προωθούν την καινοτομία. Έτσι όπως είναι σήμερα οι κανόνες, μόνο το 3% των δημοσίων δαπανών ε, περνάει το τεστ των κριτηρίων για τις δημόσιες ε, προμήθειες. Όταν αναθεωρήσουμε του χρόνου τους κανόνες, θα πρέπει να διευρύνουμε τα κριτήρια. Εγώ θα, ε, εμείς θα πρέπει να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο. Ε, όταν καθιστάς κάποια πράγματα ε, υποχρεωτικά στην πραγματικότητα, ε, δίνεις κίνητρα στους τολμηρούς, στους καινοτόμους κτλ. Αλλιώς βοηθάς αυτός που είναι τελευταίοι, οι ουραγοί. Δεν, θέλουμε, δεν πρέπει εμείς να υπερασπισόμαστε τους ουραγούς. Με αυτή την έννοια είμαι φιλελεύθερος. Έχω φιλελεύθερη λογική. ε, κάποιες, ε, κάποιες εταιρείες αναγκαστικά θα, θα εξαφανιστούν. Ε, κάπου πρέπει να είμαστε και καταστροφικά δημιουργικοί. Όταν υπερασπίζεσαι τους τελευταίους, όταν είσαι πολύ α, αμυντικός, εμποδίζεις ε, την έλευση και δημιουργία α, καινούριων παικτών. Εταιρικές σχέσεις καινοτομία. Η μόνη ανησυχία που έχω είναι ότι δεν θα πρέπει να καταστήσουμε την κρατική μηχανή, σε υπ' αυτή την έννοια, τεράστια. Αν περιμένουμε τη συνένεση 100% τίποτα θα πετύχουμε. Η κοινωνική καινοτομία για μένα είναι ο τρόπος που οργανώνουμε τη ζωή μας. Ένα άλλο θέμα η, τεχνο, η τεχνολογία συνδυάζεται εδώ με τα επιχειρηματικά μοντέλα. Και με κοινωνικές επιλογές. Δηλαδή, για μένα η κοινωνική τε... καινοτομία δεν είναι μόνο η αλλαγή της κοινωνικής ζωής, να εμπλέξουμε τον κόσμο, αλλά είναι το να εμπλέξουμε τον κόσμο ε, στην πραγματική ζωή. Ε, γι' αυτό σας καλώ όλους να είμαστε πιο τολμηροί για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Τώρα θέλω και εγώ να πω δύο φράσεις γιατί έχω πέντε, ομιλητής, πέντε ομιλητές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εισηγήτρια και δέκα λεπτά. Άρα ο καθένας θα πρέπει να είναι πιο σύντομα για να μπορούν όλοι να μιλήσουν. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είμαι ο πρώτος από τους πέντε δηλαδή. Συμφωνώ με την κυρία Μέρκες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας, να τα καταφέρουμε καλύτερα, να πλησιάσουμε περισσότερο τους πολίτες. Είναι σαφές ότι μέχρι στιγμής δυστυχώς όλα, όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα, τα πολύ διαφημισμένα, δεν έφτασαν στους πολίτες. Δεν μίλησαν στους πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά μεγάλα προγράμματα ως νέα εργαλεία, ως νέα μέσα, στο βαθμό που δεν συνοδεύονται κατά ανάγκη από τα απαραίτητα κονδύλια. Αν δούμε όλες τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν, δεκάδες είναι αυτές, ε, συχνά ε, στραγγαλίστηκαν από κανόνες και κανονισμούς. Και η αξία της έκθεσης Μέρκης θα ήταν πολύ πιο μεγάλη εάν δεν μπαίναμε σε αυτό το φαύλο κύκλο, τον παραδοσιακό. Αν προσπαθούσαμε να επικρίνουμε τη σημερινή νομοθεσία, η οποία μέχρι το 2013 θα πρέπει να προσαρμοστεί. Ισχύει για τα περιφερειακά ταμεία, για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, για μία τεράστια σειρά από μεγάλα προγράμματα, για μία πλειάδα τέτοιων προγραμμάτων. Θα πρέπει τα διάφορα μέσα και εργαλεία να συνδυαστούν περισσότερο και επίσης θα πρέπει να είμαστε και πιο έτσι, παρενετικοί, αν θέλετε. Η Επιτροπή Ίτρε όντως θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο. Ο κύριος Χατζημαρκάκης μας λέει ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά υπό το πρίσμα των περιφερειακών ταμείων. Να καταλογοποιήσουμε όλα τα ερευνητικά μέσα που έχουμε. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη και είναι καλό αυτό. Και η έκθεση θα πρέπει να το τονίζει αυτό με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Να μην μιλάμε μόνο με ευχολόγια, ε, να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Εξειδίκευση, ε, έξυπνα προγράμματα, ευφύ προγράμματα, σημαντικό. Ε, η ενιαία θηρίδα, το One Stop Shop. όλα αυτά, σύμφωνο με όλα αυτά. Το βασικό όμως είναι, στη τελική έκθεση, στην πρόταση που θα κάνετε κυρία Μέρκης, να μας πείτε με ακρίβεια τι θα πρέπει να βελτιωθεί ε, στους σημερινούς κανόνες και κανονισμούς. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Επομένως με ενδιαφέρει τα μάλλα αυτό το κείμενο. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τεράστιες αλλαγές. Γιατί ο δικός μας πολιτισμός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να ενσωματώσει με στον τρόπο ανάπτυξής του τον περιορισμένο αριθμό, την περιορισμένη ποσότητα των ε, φυσικών πόρων και το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τον αξιοποιήσουμε Καταρχάς, τη σημασία των φυσικών πόρων και το να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που ζούμε και καταναλώνουμε θα ενθαρρύνει μια νέα ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Την έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να την δούμε μέσα σε αυτό το πρίσμα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μακρόπνοα την έρευνα και ανάπτυξη. Μέσα σε ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα. Η δουλειά που κάνουν όλες οι επιτροπές που γνωμοδοτούν επί της έκθεσης αυτής είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει η κοινωνία μας ε, να αλλάξει τον τρόπο που ζει, τον τρόπο που σκέφτεται. Ευχαριστώ την, κυρία Μέρκες για τα σχόλια της και την παρουσίαση. Ευχαριστώ την ε, ανακοίνωση της ε, Επιτροπής για την ε, καινοτομία. Είναι καλό κείμενο. Λέει πολλά πράγματα και για άλλα θέματα, εκπαίδευση κτλ. Συμφωνώ με τον ορισμό της καινοτομία, Μίλησαμε για την κοινωνική καινοτομία, Η περιφερειακή καινοτομία είναι πολύ σημαντική επίσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει και μια θεσμική καινοτομία, ιδίως ε, στις ε, κρατικές, ε, στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό, δεδομένης της κρίσης σήμερα, να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτό. Το κείμενο θα πρέπει να εξισορροπηθεί περισσότερο. Να μιλήσουμε πιο ισορροπημένα για τα διάφορα είδη καινοτομία. Να δώσω μεγαλύτερη έμφαση και στην βιομηχανική καινοτομία. Η Ένωση Καινοτομία είναι σημαντικό για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας ε, παγκόσμια για να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και να διατηρήσουμε το ρόλο μας, ε, τον εξαγωγικό, ε, στις παγκόσμιες αγορές. Και ενώ σε βιομηχανικούς τομείς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε για να αναγεννηθούν. Αλλά το θέμα είναι να κατακτήσουμε και την ηγετική θέση παγκόσμια. Αν δείτε τον ε, πίνακα βαθμολογίας για τη βιομηχανία που ετοίμασε η Κομισιόν, ε, ο πρώτος τομέας είναι η βιομηχανία και η αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτούς τους τομείς ε, στα πλαίσια των πόρων που έχουμε, ούτως ώστε ε, να χρησιμοποιούμε με αποτελεσματικό τρόπο τους πόρους μας και να διατηρήσουμε τον ηγετικό ρόλο παγκόσμια. Εξαγωγικό ηγετικό ρόλο. Συγχωρείτε, χάσαμε την κυρία Σαρτόρη που ήταν η συγγήτρια. Της δίνω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδη συγγήτρια του ΕΛΚΑ και ω τέτοια συμμετείχα στη συνεδρίαση τη 24 η Νοεμβρίου με την εισηγήτρια και συμμερίσομαι τα όσα είπαν και άλλοι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα ότι και η δουλειά που έκανε και η συγγήτρια αλλά και η Επιτροπή μας είναι καλή δουλειά και προς κατεύθυνση. Εγώ τώρα έχω την πρόθεση να σταθώ σε κάποια σημεία που θεωρώ πιο σημαντικά. Καταρχάς, και το θέμα της καινοτομίας, όπως έχει υποθεί και στο παρελθόν, για άλλα σημαντικά θέματα να γίνει οριζόντιο θέμα, να ενσωματωθεί σε όλους τους κανονισμούς, σε όλες τις οδηγίες που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της ε, οριζόντιας ε, ενσωμάτωσης ε, της Δεν έχει να λέμε «Α, καινοτομία και εδώ, καινοτομία και εκεί, καινοτομία και παραπέρα». Από σήμερα και στο εξής, ό,τι κάνει η Ευρώπη θα πρέπει να έχει και μια διάσταση καινοτομία. Αυτό είναι το πρώτο. Κάτι άλλο. Δεν θέλω να επανερχόμαστε στο παρελθόν, σε αυτά που κάναμε ήδη. Στο πρόγραμμα έρευνας ε, που αφορά την ε, δημόσια διοίκηση. Κάτι άλλο που με βρίσκει σύμφωνη είναι αυτή η ενιαία θηρίδα προς την οποία μπορούμε να απευθυνθούμε. Αυτό το θέμα συνδέεται με την απογραφειοκρατικοποίηση, που είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχει η Ένωση. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την δομή για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο περίπλοκο και γραφειοκρατικό κόσμο όπως αυτός της Ένωσης. Η προπαρασκευαστική δουλειά θα πρέπει να γίνει εδώ και να τους δώσουμε αυτή την ενιαία θηρίδα προς την οποία να μπορούν να απευθυνθούν. Ε, πρώτο τελευταίο σημείο. Η Ευρώπη θα πρέπει να θέσει εαυτόν το στόχο όχι μόνο να βοηθήσει και να υπερασπιστεί την, τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, αλλά να τα κάνει και γνωστά. Είναι άπειρε οι καινοτομίε, άπειρα τα διπλώματα ε, ευρεσιτεχνία που έχουν κατατεθεί, αλλά δεν τα ξέρει κανένας. Το κοινό δεν τα ξέρει. Και επομένω δεν χρησιμοποιούνται αυτέ οι καινοτομίε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ακόμα, αλλά ας πω ακόμα ένα μόνο. Απευθύνομαι στους συναδέλφους και όχι στον πρόεδρο. Κύριοι συνάδελφοι, ας είμαστε λιγότερο φιλοσοφικοί, δεν χρειάζεται να θεωρητικολογούμε τόσο πολύ, έτσι. Ορισμένοι από αυτούς που μίλησαν, ε, που μέσα έχουν φύγει και όλα, ήταν πάρα πολύ φιλοσοφικοί. Κρατικές συμβάσεις, διαγωνισμοί στο δημόσιο. Όταν μιλάμε για τους διαγωνισμούς, θα πρέπει να βάλουμε κάποια δεσμευτικά στοιχεία. Δεν θέλω να μιλήσω για τη σχετική οδηγία τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο ακόμα θα πρέπει να εντάξουμε την καινοτομία. Όπως σας είπα, να την αντιμετωπίσουμε οριζόντια. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στα μοντέρνα και γνωστά σημεία, που είναι σημαντικά, όπως είναι η ενέργεια και γενικά τα πράσινα θέματα. Να ξεπεράσουμε μόνο, να ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά ασφάλεια, υγεία, καινοτομία και στην ασφάλεια και καινοτομία και στην υγεία ε, και στους διαγωνισμούς στο δημόσιο παντού, καινοτομία παντού. Αυτά λοιπόν από, το, από την ε, πολιτική μου ομάδα θα συνεχιστεί η δουλειά και θα πλαισιώσουμε για να βοηθήσουμε την εισηγήτρια και εμείς όσο μπορούμε. Ο κύριος Ούντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπάρξουν ορισμοί. Μιλάμε για έρευνα και καινοτομία. Τι είναι η έρευνα, τι είναι η καινοτομία. Ο, <laughs> ε, ο Σενάδο Ντεγκόλ έλεγε ότι έχουμε πολλούς ερευνητές, αλλά κάποιοι ε, θα πρέπει να βρίσκουν κιόλας, όχι μόνο να ψάχνουν. Επομένως, ορισμοί. Λείπει επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για την καινοτομία στο περιβάλλον. Μιλήσαμε για καινοτομία στη βιομηχανία, στην οικονομία, ε, για την κοινωνική καινοτομία μιλήσαμε επίσης ένα θαυμάσιο κεφάλαιο, αλλά λείπει αυτό το κεφάλαιο. Και όπως είπε και ο συνάδελφος πρώτη, που να μιλάει επίσης και για την έλλειψη πόρων. Επίσης μιλάμε για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα. Εγώ ανήκω σε ένα κράτος μέλος όπου η διοίκησή του έχει, έχει κάνει πολλές καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση προσοχή σε αυτό το θέμα. Να διακρίνουμε λοιπόν αυτή την καινοτομία από τις υπόλοιπε. Τελευταία παρατήρηση για την εισηγήτρια, η σχέση με τα κράτη-μέλη τα, στη σύνοψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέσσερα σημεία μιλάμε για τη σχέση με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εμπλέξουμε το συντομότερο δυνατόν και τους εθνικούς βουλευτές, ούτως ώστε η σχέση Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, για αυτό μεγάλο θέμα, να μην ε, δημιουργεί αποκλήσεις στις απόψεις μας. Επίσης, οι τοπικές ε, κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις μάλλον, και οι τοπικές κυβερνήσεις ε, ενδιαφέρονται πολύ για αυτό το θέμα. Να λάβουμε υπόψη μας και την Επιτροπή των Περιφερειών και την απόψή της. Herzog. We have seen... Στα γρήγορα να σας πω ότι στη συζήτηση περί περιπολογισμού είδαμε πως διστάζουν ιδιαίτερα τα μέλη του Συμβουλίου να στηρίξουν την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ίδιο σημαίνει και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε πως ε, το αδύνατο σκέλος των κυβερνητικών προγραμμάτων είναι η καινοτομία. Θέλω λοιπόν μια πολύ στεναρή διατύπωση έτσι ώστε να φαίνεται αυτό, γιατί βέβαια η καινοτομία μέσω της συνθήκη Λισαβόνα είναι πλέον υποχρεωτική. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης των επιδόσεων των εθνικών κυβερνήσεων και νομίζω πως θα πρέπει η δράση τους να βαθμολογείται και να ξέρουμε σε ποιο βαθμό είναι επιτυχημένη. Δεν μπορούμε να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα, δεν θα έχει ε, εργαλείο χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά παράλληλα να μην εξασφαλίζουμε ότι τουλάχιστον τα όσα γίνονται με εθνική χρηματοδότηση θα μπορούν κάπως να υπολογιστούν. Παρακαλώ λοιπόν κάτι, ένας τρόπος υπολογισμού να ενταχθεί. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε κάτι να πείτε, αν καταφέρετε να είστε σύντομος θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω πως βιάζεστε. Να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια, την κυρία Μέρκης, για πολύ καλή δουλειά και να σας πω πως ακόμα και τα όσα άκουσα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και από όλους τους κοιόδης εισηγητές. Απλώς δεν θα προλάβω τώρα να τα σχολιάσω. Το μόνο που θα πω εδώ είναι ότι και εμείς συμφωνούμε πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Διαφορετικά η επίγουσα κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει η καινοτομία δεν θα ξεπεραστεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ενσωματώσουμε ε, στις διάφορες πολιτικές μας, περιφερειακή πολιτική, στην υγεία, ε, το σκέλος της καινοτομίας. Αν φανούμε φιλόδοξοι, θα πρέπει να το κάνουμε με έναν ευφυή τρόπο και να κάνουμε μια ευφυή ε, δημοσιονομική ολοκλήρωση. Δηλαδή, να είμαστε σίγουροι πως δεν υποσκάπτουμε το μέλλον μας με λήψη βιαστικών αποφάσεων δεδομένης της κατάστασης μέσα στην οποία ζούμε. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα θέμα το οποίο, οι δημόσιε προμήθειες, με είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και καιρό την Κομισιόν. Θεωρούμε πως οι δημόσιες προμήθειες έχουν ένα τεράστιο δυναμικό, το οποίο εμεί θα πρέπει να εξερευνήσουμε για να δούμε κατά πόσο εκεί μπορούμε να εντάξουμε την καινοτομία. Να διαβεβαιώσω την κυρία Μέρκης που εξέφρασε κάποιες ε, αμφιβολίες για τις εταιρικές σχέσεις στην καινοτομία. Να σας πω πως γίνεται αυτή τη στιγμή μία πειραματική εφαρμογή του Healthy Aging και ελπίζουμε σε αυτό να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο όσο δραστήρια γίνεται, γιατί αυτό θα εξηγήσει και πώς τα εταιρικά αυτά σχήματα θα τα διαχειριστούμε, τι παραδοτέα ε, περιμένουμε. Και παρακαλώ πολύ, ε, θέλουμε τη δική σας εμπλοκή στο πειραματικό αυτό σχέδιο. για να κάνουμε κάποιε προσπάθειε οι οποίε θα λάβουν υπόψη, κατά όσο είπε ο κύριο Χατζημαρκάκη. Ναι, όντω θα πρέπει να δίδονται κάποια μπόνου και με χαρά θα ακούσω τις απόψει στο σημείο αυτό. Ένα σημείο μόνο ξέχασα για τι εταιρικέ σχέσεις. Η κυρία Μέρκη το έθιξε. Δεν είναι νέα μέσα αυτές οι εταιρικέ σχέσεις δεν αποτελούν νέες πηγές χρηματοδότησης. Είναι μια διαδικασία ή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εντάξουμε αυτή την ολοκληρωμένη διαδικασία στην οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί σας εσύ. Καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας της κοινοτομίας, από πρώτη ιδέα μέχρι τη χάραξη προτύπων, μέχρι τη βαραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες των πολιτών. Δεν είναι ένα νέο μέσο, υπάρχει εδώ και καιρό. Καταλαβαίνω βεβαίως ε, τις ε, δυσκολίες σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ για τα σύντομα αυτά σχόλια και δεν ξέρω αν η κυρία Μέρκης θέλει κάτι να πει ακόμη ή αν θα ήθελε, αλλά παρακαλώ σύντομα. Briefly react. So much has been said. Θα είμαι πολύ σύντομη. Βεβαίως, ε, Βεβαίως θα πρέπει να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Στόχος μας τα αστέρια, αλλά αν μόνο φτάσουμε στο φεγγάρι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μου είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι. Ναι, ε, συμφωνώ. Αλλά εμένα η στάση μου δεν θα, δεν θα είναι αμυντική στο σημείο αυτό. Θα σας πω που συμφωνώ, ας είμαστε, δεν θα πω επιθετικοί, αλλά είμαστε, ας είμαστε τουλάχιστον ε, πρόθυμοι να φτάσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε για να πετύχουμε κάποια κέντρα αριστείας και χαίρομαι που η Επιτροπή Πολιτισμού γνωμοδότησε γιατί πιστεύω πως όλα τα μέσα θα μας βοηθήσουν και ανησυχώ ανησυχώ που η καινοτομία δεν μοιάζει να ευθυγραμμίζεται με τις ε, κοινωνικές επιταγές τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν να εντάξουμε παντού την καινοτομία, πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με τις πολιτικές σε άλλους χώρους και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όλα τα εργαλεία θα δουλέψουν υπέρ της καινοτομία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Βέβαια, οι κυβερνήσεις, το είπα και εγώ, είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δημόσιες προμήθειες λοιπόν είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Ξέρω πως υπάρχουν και άλλες επιτροπές που θέλουν να γνωμοδοτήσουν. Θα καταφέρουμε όμως να είμαστε ανοιχτοί. Θα μιλήσουμε με την ΕΜΚΟ και για την εσωτερική αγορά και για τις δημόσιες προμήθειες και για τη χρηματοδότηση. Το συζητάμε και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία και να σχεδιάσουμε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα. Αυτή η ένωση της καινοτομίας θέλει να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και επιταγές και βέβαια καταλαβαίνετε πως η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πρώτες προκλήσεις που θα πρέπει να μας ανησυχούν. Να επιθυμίσω άλλωστε στους συναδέλφους πως στο ψήφισμά μας εμείς ξεκαθαρίσαμε πως η ευφυής χρήση των πόρων είναι η βασική αρχή για οποιαδήποτε εταιρική σχέση καινοτομίας. Άρα λοιπόν εκεί θα στρέψουμε και τα βέλη μας και με χαρά έχω σκοπό να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για τα σχόλια που έκαναν και για τα θέματα που σε απασχολούν και με τα περισσότερα από τα οποία συμφωνώ. Ευχαριστώ που ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό της ημερησίας διατάξεως και προχωρούμε γρήγορα στην ε, ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, οπότε κάνουμε την ε, πρώτη ψηφοφορία για την έκθεση Μαρινέσκου σχετικά με την ε, χρηματοδότηση της καινοτομίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακαλώ πάρτε τον κατάλογο ψηφοφοριών μπροστά σας. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές Με συγχωρείτε, με πήρα άλλη, ένα άλλο κατάλογο ψηφοφορίες, ε, ε, χωριστή ψηφοφορία, ένα υπέρ κατά αποχές, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος για την 8. Ε, Λίγοι, Απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, το 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 15. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Τώρα, συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και παραμένει τώρα... Το δεύτερο μέρος της 32 υπέρ. Κατά. Ποιο δεύτερο μέρος. Εφόσον ποιος είναι υπέρ της, ε, του 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα στην 24 υπάρχει μία προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές αποφασίζεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά ελέγχουμε το δεύτερο μέρος της 23. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ε, το ΕΛΚ έχει ένα παραπάνω, όχι. Ένα παραπάνω έχει το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα. Και εγκρίνεται. Τώρα στην 26 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές 28 ε, ε, υπέρ. Κατά αποχές αποφασίζεται. 30 υπέρ. Όχι. Είμαι πιο γρήγορος από όλους λέει ο εισηγητής. Τώρα 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές αποφασίζεται. 34 υπέρ. Είμαστε στην 34. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 τώρα σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα της 35 υπέρ κατά αποχές αποφασίζεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά Ελέγχουμε την 36 ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απερίφθη. 40. Κύριε Ζαντό. Θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι έχει ισχύσει η 38 με την προφορική τροπολογία, δεν την αναφέρατε. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία. Αναφέρεται στον κατάλογο. Εγώ στον κατάλογο μου στο 38 δεν βλέπω προφορική τροπολογία, λέει ο πρόεδρος. να το διαβάσω. Όχι, ε, τώρα μου είπαν ότι άργησε να υποβληθεί η προφορική τροπολογία. Η άλλη... Με συγχωρείτε, εγώ φώναξα για το 38 δεν αναφέρθηκα για, στην προφορική τροπολογία, αλλά αυτό ήταν δικό μου λάθος, αλλά κανείς δεν μου το ανάφερε. Θέλετε να, να ε, επαναλάβουμε με την προφορική τροπολογία, κύριε Τσίτσεστερ. Ναι κύριε Πρόεδρε, την έχουμε ελέγξει την προφορική τροπολογία. Τότε δηλαδή δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει. Δηλαδή, εφόσον μία ομάδα απορρίπτει την προφορική τροπολογία και απερίφθηκε 37, τώρα πάμε στην 40 χωρίς προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της 40 χωρίς προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 41. Θα ελέγξουμε τη 40 χωρίς την προφορική τροπολογία παρακαλώ. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα του 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τώρα ερχόμαστε σε δύο χωριστές ε, ψηφοφορίες. Το 42 έχει δύο φορές split vote. Μπορούσαμε να κάνουμε τέσσερα στη σειρά και όχι δύο επί δύο. Από την πρώτη split vote το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο Δεύτερο split vote, πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην ε, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία ξεκινά. Λίγη. και εγκρίθηκε. Ε, συγχαίρω ε, τον εισηγητή. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα, στο 9, αλλά ο κύριος Τούρμες ε, θέλει καταρχήν διαδικατηρικό. Την προφορική τροπολογία. Ο Τσάλς δεν έχει και πολύ όρεξη σήμερα, δεν μπορέσαμε να την ψηφίσουμε λοιπόν. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τους εσωτερικούς μας κανόνες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στη συνάντηση των συντονιστών τον Ιανουάριο τι γίνεται με την προφορική τροπολογία. Ε, Ποιο είναι ο κανόνα για την προφορική τροπολογία. Δεν τα ξέρει και η γραμματεία τελικά τι γίνεται. Αυτό ήταν ένα δικό μου λάθος όπως είπα και μετά το αναθεώρησε. Μπορεί κανείς να υποβάλει κατά την διαδικασία μία προφορική τροπολογία αλλά ε, όταν ένας θα απορρίψει ε, λύγει το θέμα. Τώρα πάμε στην ψηφοφορία του σημείου 9. Ε, ο εισηγητής δεν έχει πολλά να πει και πάμε κατευθείαν στη συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται για την έκθεση 2010. Ε, δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ. Έξι. Λοιπόν, με συγχωρείτε πρώτα, η έξι λέει ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της έξι. Υπέρ της έξι. Κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 υπέρ κατά αποχές απερι, ε, ε, 14 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 4 ποιος είναι υπέρ κατά Αποχές εγκρίθηκε. 16 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος. Με συγχωρείτε με συγχωρείτε, το πρώτο, ε, ε, το πρώτο τμήμα καλύφθηκε από τη συμβαστική 4, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές αποφασίστηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απεφασίστηκε, εγκρίθηκε επίσης. Ερχόμαστε τώρα στο 20 υπέρ. Κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 20. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Και πάλι το έλκα ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος στις 22 ξεκινά λίγη απερίφθη. Ας ξαναξεκινήσουμε. 22, ε, ξεκινά για την 22 πάλι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. Απερίφθη. Η 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 25. Υπέρ κατά αποχές αποφασίστηκε. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Ε, συμβιβαστική 6. Έλεγχος της 28, ευχαρίστως, ηλεκτρονικός έλεγχος της 28, ξεκινά, λίγη, Ναι, ε, μικρή ε, λέει πλειοψηφία. 6 υπέρ κατά αποχές. Αποφασίστηκε 30 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε 32 ε, χωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απερίφθη επίσης 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινά. Λίγη. Και το τελικό αποτέλεσμα ε, εγκρίθηκε. Συγχαίρω ήταν η τελευταία ψηφοφορία πριν από τα Χριστούγεννα σημαντικό γεγονός ε, χαίρομαι για την συνεργασία αλλά κύριε Λάνιε εάν είστε τόσο ευγενικός θα κάνουμε δύο έκτακτες συνεδριάσεις δεν τέλειωσε όμως η συνεδρίαση τώρα έχουμε ακόμη συζητήσεις οπότε δεν υπάρχει λόγος να φύγετε και τώρα είμαστε στο σημείο 10 όπου πρόκειται για τις σχέσεις ε, μεταξύ ΕΕ και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Καταρχήν έχει μόνη της και αποκλειστικά το λόγο Παρακαλώ συνάδελφοι, αν θέλετε να συζητήσετε εκτός εθούσης, αν θέλετε να φύγετε αποχωρήστε γρήγορα, αλλά μην διαταράσετε τη συνεδρίαση. Also immer, immer mündlich. Ich habe da nur einen Fehler gemacht. Als sie sagt, es ist zu spät, da habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich besser Mund gehalten. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να περιμένουμε δύο λεφτά ακόμη μέχρι να ηρεμήσουν. It is, it possible? Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, κύριε Μπρεζίνα, ε, κύριε Βινταλκουάντρας και ορισμένοι άλλοι, μπορείτε να σταματήσετε τα πηγαδάκια και να έχουμε ε, χρόνο για να γίνει η επίσημη συζήτηση. Όχι. Bye bye. No, is not necessary. It's the form of discipline. They come too late, they talk,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 Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τώρα μπορώ να ξεκινήσω, ε, διότι και εγώ τέλειωσα τη συζήτησή μου και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σας παρουσιάζω εδώ την τοποθέτησή μου σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις, ε, ε, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και είμαι πολύ ευγνώμων διότι αποφάσισε η ε, Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων να ε, καταρτήσουμε μία έκθεση με αποκλειστικό θέμα της σχέσης ε, με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου γιατί αυτό, αυτή η περιοχή για μας είναι μία στρατηγικά πολύ σημαντική περιοχή και χαίρομαι ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μας έδωσε αυτή την εφορία να παρουσιάσουμε σχολιάσουμε τρία θέματα τα οποία μας καλύπτουν και να περιληφθεί στην τελική έκθεση και η δικιά μας γνωμοδότηση. Ε, έχω καταρτήσει ένα έγγραφο όπου αναφέρομαι εις την συνεργασία με τις χώρες του κόλπου καταρχήν σχετικά με την ενέργεια, δεύτερον σχετικά με τη βιομηχανία και ιδίως πρώτες ύλες και τρίτον ε, καινοτομία. Καταρχήν όσον αφορά την ενέργεια. Νομίζω ότι τα ορυκτά καύσιμα τα οποία βρίσκουμε ε, αποτελούν ε, την πιο σημαντική πηγή καυσίμων για την Ευρώπη για να καλύψει τις ανάγκες της και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε στενή επαφή με τις χώρες που μας προμηθεύουν και χαιρετίζω την Joint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 αναφέρονται οι στατιστικές για την παραγωγή πετρελαίου με περισσότερη διαφάνεια. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργείας υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες για το υγροποιημένο αέριο και ε, το φυσικό αέριο και γι' αυτό όσον αφορά την Αραβική Χερσόνησο την επισκέφτηκα προ λίγων μηνών πήγαμε και στο Κατάρ και εκεί είδαμε ε, την τεράστια πλατφόρμα η οποία έχει κατασκευαστεί ε, πριν από 10 χρόνια για να υγροποιεί το αέριο και να το εξάγει και το ερώτημα είναι αν εδώ υπάρχει ε, μία πύλη υποδοχής για τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο και αυτό το σημείο το έχω περιλάβει στην έκθεσή μου όσον αφορά το υγροποιημένο αέριο, το LNG δηλαδή, ε, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει αυτή η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βεβαίως αναφέρομαι και στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και ε, τη συνεργασία μας την οποία πρέπει να εντείνουμε όσον αφορά την αιωλική και ηλιακή ενέργεια και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες εις, ε, να επενδύσουμε περισσότερο εις ε, τις ενέργειες αυτές. Αυτή είναι η, μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική για τους Ευρωπαίους. Πιστεύω ότι και για τη βιομηχανία χρειάζεται μια σύσφυξη των σχέσεων στον τομέα αυτό και πολιτικά χρειάζονται δύο πράγματα. Καταρχάς να καταργηθούν ε, τα οι εμπορικοί φραγμοί που υπάρχουν ακόμη και ε, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου την οποία διαπραγματευόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, δεν έχει ακόμη τελεσφορήσει και πιστεύω ότι στη γνωμοδότηση είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ε, για να τελεσφορήσει. Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και καινοτομίας, θα ήθελα εδώ να σας πω ποιες είναι οι εμπειρίες μας. Ο κύριος Ρούμπικ που ήταν μαζί στο ταξίδι, ε, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι δυνατότητες υπάρχουν για τους ε, ε, φοιτητές στην περιοχή. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν ή στο πρόγραμμα Erasmus Mundus παραδείγματος χάρη, αλλά εκεί σε αυτές τις χώρες δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες οπότε πρέπει να προωθήσουμε το ότι μπορούμε να προσφέρουμε από πλευράς Ευρώπης και ιδίω όσον αφορά τους ξένους φοιτητέ να τους καλέσουμε να έρθουν στην Ευρώπη να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας να επενδύσουμε στον τομέα αυτό και όπως σας ε, είπα στην έκθεσή μου τονίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουμε γνωστοί εις ε, τα πανεπιστήμια να υπάρχει μία στενότερη συνεργασία σχετικά με την τεχνολογία διότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να προωθήσουμε και στο Energy Park του Κατάρ παραδείγματος χάρη αλλά η Ευρώπη δεν έχει μία ισχυρή παρουσία στην περιοχή αυτή και θα ήταν σκόπιμο να την ενισχύσουμε. Το τελικό πιο μεγάλο πρόβλημα σαν Ευρωπαίοι που αντιμετωπίζουμε εκεί είναι ότι έχουμε μία μόνο εκπροσώπηση στη Σαουδική Αραβία για όλη την περιοχή. Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγάλος αδερφός των μικροτέρων χωρών, ο Μαν, Μπαχρέιν κτλ. Και, και θα ήταν σκόπιμο να προσπαθήσουμε και στις άλλες μικρότερες αλλά για μας ε, τους Ευρωπαίους στρατηγικά τόσο σημαντικές χώρες να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση και ελπίζω ότι θα περιληφθεί στην έκθεση και ότι θα συνενέσει και η ηγετική επιτροπή. Τέλος αναφέρουμε στην στενή συνεργασία με τις ε, χώρες του κόλπου όσον αφορά την ε, ενέργεια, την ασφάλεια ασφάλεια πρώτων υλών και την καινοτομία. Θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν και θα παρακαλούσα να στηρίξετε τις προτάσεις μου, αλλά βέβαια είμαι ανοιχτή σε προτάσεις οποίες ενδεχομένως θέλετε να μου διατυπώσετε. Ευχαριστώ. Θέλουν οι πολυάριθμοι ε, σκιώδεις συγητές να παρέμβουν. Εδώ βλέπω θα παρέμβει ο μη σκιώδης ε, εισηγητής. Θέλω να ευχαριστήσω την Αγγέλικα Νίμπλερ η οποία οποία ηγήθηκε της αντιπροσωπείας και ε, μας δείχνει η έκθεση αυτή πολύ καλά αν να επιτύχουμε. Πρέπει να αυξήσουμε την εκπροσώπησή μας στις χώρες του κόλπου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σκόπιμο θα ήταν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε. Δηλαδή σε κάθε μία από τις ε, χώρες αυτές καλό θα ήταν να έχουμε μία πρεσβεία και θα μπορέσει ίσως ε, να βοηθήσει και σε οικονομίες για τις χώρες αυτές οι οποίες τώρα χρειάζεται να εκπροσωπούνται και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ανώσεως και θα βελτιώσει τη συνεργασία. Το διοξίδιο του άνθρακος είναι σημαντικό θέμα ή στην παραγωγή αερίου και πετρελαίου και γι' αυτό οι μειώσεις του διοξιδίου του άνθρακος όχι μόνο στην αποθήκευση αλλά και για τα χημικά καύσιμα, chemical fuel, θα πρέπει να μειωθούν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Scientific Options Assessment τόνισε ότι το διοξίδιο του άνθρακος ή ε, τα chemical fuel πρέπει να εξεταστεί και να δούμε πόσο ε, το διοξίδιο του άνθρακος μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ή στις βιομηχανικές ε, διεργασίες και να εφαρμοστεί. Δύο θέματα κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά κατήρχας ε, το European Research Council και ε, οι υποτροφίες οι οποίες δίδονται και οι οποίες είναι σημαντικές ε, και για τα κράτη αυτά και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Ουγγαρία θα μπορούσε να συνεργαστεί καλύτερα με, τις, με τα πανεπιστήμια της περιοχής. Αρχή, Δεκεμβρίου υπάρχει το Oil Show στο Κατάρ όπου εκπροσωπούνται όλοι οι πάροχοι πετρελαίου και αερίου και καλό θα ήταν ίσως ε, ε, η τροπή μας να επισκεφθεί κάποτε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι δεν βλέπω κανείς να ζητά τον λόγο οπότε η έκθεση είναι τόσο καλή ώστε κανείς δεν χρειάζεται να τη σχολιάσει και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Κυρία Νίμπλερ, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, σχετικά με τον συνάδελφο Ρούμπιχ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις προτάσεις. Αντιλαμβάνουμε ότι θα κάνει τροπολογίες για πράγματα τα οποία δεν έχω θίξει και καλό θα ήταν εάν ε, γίνει αυτό το oil show στο Κατάρ να στείλουμε κάποιον ε, εγώ πάω αν θέλετε αλλά αν κάποιος ενδιαφέρεται νομίζω ότι δεν θα ήταν κακό για πλευράς ενεργειακής ασφαλείας και θα ήταν σκόπιμο να το εξετάσουμε κύριε Πρόεδρε αν υπάρχουν οι δυνατότητες να υπάρξει μία επίσημη εκπροσώπησή μας ε, και θα πρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα γιατί είναι κάτι που γίνεται, α με συγχωρείτε, όχι την άλλη εβδομάδα, του χρόνου. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να το περιλάβετε στις συζητήσεις σας κατά τρόπον ώστε να ε, ε, πάει ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής μας αλλά με κάποια προσωπικότητα. Νομίζω ότι μεταξύ μας λύσαμε το θέμα. Ωραία. Σημειώνουμε τότε αυτή την, ε, αυτό το θέμα. Ξέρετε την προσθεσμία για τις τροπολογίες, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Θέλετε κάτι να πείτε. 8 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τις ε, ε, τροπολογίες. Δηλαδή όποιος θέλει να κάνει κάτι θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα πριν τα Χριστούγεννα. Έκλεισε το μικρόφωνο του Προέδρου. Λοιπόν, εδώ αναφερόμαστε στον ε, τουριστικό προορισμό αναψυχής και δίνω τον λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη. Ε, ε, όποιος, όποιος σκέφτεται διακοπές καλά κάνει γιατί πλησιάζουν οι διακοπές. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα του τουρισμού Ίσως θα εκπλήσει ορισμένους ότι το συζητάμε στην Επιτροπή μας Ήτρε, αλλά ε, ε, μη, ε, ένας, ένας επίτροπος, ο κύριος Ταγιάννη, το έθεσε στην ημερήσια διάταξη και αυτό για κάποιο σωστό λόγο, διότι ο τουρισμός περιλαμβάνεται από τις συνθήκες της Λισαβόνας εις τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν υπάρχει υπεύθυνη αρχή για τον τουρισμό βέβαια στηρίζουν τα κράτη την ε, δραστηριότητα αυτή αλλά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός του κόσμου και ο τουρισμός είναι η τρίτη κοινωνικο-οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφτασε λοιπόν η ώρα να το αντιληφθούμε και ότι τουρισμός όπως και οι άνθρωποι στις κοινωνίες μας αλλάζει και ε, πρέπει να προσαρμοστούμε. Άρα εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να κοιτάξουμε και ενδεχομένως να κατακρίνουμε τις κινήσεις οι οποίες γίνονται διότι υπάρχουν ερευνητές ε, οι οποίοι ε, πλέον πλέον είναι ε, ε, μουσιακοί και ίσως μουσιακά ενδιαφέρουν τον, τους τουρίστες. Αλλά ε, πρέπει να πούμε ότι από πλευρά αριθμών βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται προς την Ευρώπη και ε, ιδίω από την Βραζιλία, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία και οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται ηλικιωδώς. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ε, μια τουριστική βιομηχανία διότι πολλές ε, επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες στον τομέα αυτό και είναι ε, ένα προσόν το οποίο έχουμε αντιληφθεί είμαστε ο πιο ενδιαφέρον προορισμός με την ιστορία μας και τη γεωγραφική μας θέση και από πλευράς εσωτερικής αγοράς για την πολιτική εσωτερικής αγοράς έχουμε μια αξιόπιστη βάση την οποία έχουμε δημιουργήσει. Είναι ενδιαφέρον παραδείγματο χάρη να, να κινηθεί κανείς από ότι την Ολλανδία προς ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσης να έχει περισσότερο ήλιο αλλά και αξιόπιστες τουριστικές υπηρεσίες. Εάν θέλουμε όμως να θέσουμε ε, νέα βάση στον τουρισμό πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να συμβουλεύσουμε στην τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης για να βελτιωθεί και εδώ βλέπω πολλά σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Η γαστρονομία όπου θεωρούμε ότι η διατροφή είναι σημαντική για μια υγιεινή ζωή οπότε και στη γαστρονομία υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα οδηγήσουν σε μια βελτίωση της ποιότητος. Βλέπουμε τη δημογραφική αλλαγή ε, για τον πραγματικό τουρισμό. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι αλλά οι οποίοι ταξιδεύουν. Άρα αυτό το θέμα είναι ενδιαφέρον και αν το συνδυάσουμε με το προηγούμενο μπορούμε να προκαλέσουμε πολλές καινοτομίες όπως είπαμε σήμερα το πρωί και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε αυτή την συνεργασία καινοτομία ε, για να έχει κανείς περισσότερα χρόνια ε, ζωής με ψηλή ποιότητα. Χρειαζόμαστε επίσης μία, ε, μία ενοποίηση των κανόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη διότι στον τουρισμό νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τις χώρες της Μεσογείου που είναι τοριστικοί προορισμοί διότι όλοι τώρα πλέον θεωρούμε ότι οι ε, δραστηριότητες μας ε, για να είμαστε υγιείς εξασκούνται κατά τον ελεύθερο χρόνο τα check-up παραδείγματος χάρη η ιατρική έλεγχη οι οποίοι ε, δεν πρέπει να γίνουν ίσως ανά ανάμεσα σε δύο συνεδριάσεις ε, ήτρε ε, όπου ε, δημιουργούν ένταση αλλά μπορεί να πάει διακοπές στην Κρήτη, στην Σικελία, στην Αυστρία να κλείσει διακοπές για δύο εβδομάδες εκ των οποίων τέσσερις ημέρες θα αφιερώσει για μια ιατρική εξέταση, ένα check-up. Ίσως ήθελε να κάνει κάνει και μία μικροεπέμβαση την οποία θα συνδυάσει ε, με τις διακοπές του ε, αυτά τα οποία λέτε τώρα είναι προστασία δεδομένων και ίσως θα σου χυμίξουν οι συνάδελφοι. Εντάξει, ε, τότε θα είναι ε, διάφορες διακοπές προς την Αυστρία, προς την Κρήτη και πιο διαρκείας παραμονές. Αλλά μπορούμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες τις ξενοδοχειακές με τις υγειονομικές και σε αυτή την Επιτροπή ε, έχουμε επέμβει με την δεύτερη ε, οδηγία για την ε, κινητικότητα των ασθενών και αυτά θα είναι δραστηριότητες που θα πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν δηλαδή νέες δυνατότητες ώστε ο τουρισμός να προωθηθεί. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε μία σφραγίδα ποιότητος. Έχουμε ε, τις ε, μπλε σημαίες για το, τη θάλασσα ε, που μας δείχνει ότι η θάλασσα είναι καθαρή και οι ακτές ποιοτικέ, θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε μπλε σταυρούς όπου θα υπάρχει υψηλότερη βαθμολόγηση όταν υπάρχει ιατρικό κέντρο ενδεχομένως μέσα στο ξενοδοχείο και οπότε όποιος έχει τρεις σταυρούς θα είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Ξέρουμε λοιπόν ότι, όλη, ε, ε, η αγορά για την ε, ιδιωτική περίθαλψη στο μέλλον αυξάνεται πάρα πολύ, έχει δηλαδή πολλές δυνατότητες αρκεί να δημιουργηθούν αυτά τα ποιοτικά κριτήρια και οι επίτροποι Νταγιάννη και Ντάλι ήδη έχουν σκεφτεί το θέμα αυτό αλλά ίσως και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε χρήσιμες ιδέες και αυτό αυτό προτείνω. Υπάρχει και ένας αρνητικός τομέας που είναι η, ε, η οδική κυκλοφορία διότι βλέπουμε ότι οι 25.000 ε, τουρίστες πλήττονται από οδικά ατυχήματα και ε, στον τουρισμό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και σε προβλήματα οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ενιαία δεν υπάρχουν νέοι κανόνες και ε, παραδείγματος χάρη είναι ε, ε, το, το Βέλγιο υπάρχει προτεραιότητα από δεξιά προς αριστερά πράγμα το οποίο ίσως δεν ισχύει στην Ιταλία ή στην Ελλάδα πρέπει να, υπάρχει ενιαία, να υπάρχουν ενιαία χρώματα ενιαίος τρόπος σημάνσεως των ταξί κατά τρόπο ώστε ε, να μειώσουμε όσο δυνατόν τους κινδύνους στις οδικές μεταφορές. Θα ήμουν ευτυχής εάν αυτή η γνωμοδότηση ε, μπορεί να υιοθετηθεί από τους συναδέλφους, ε, θα μπορέσουν να σχολιάσουν και να μου δώσουν επιπλέον ιδέες. Τον Ιανουάριο θα παρουσιάσουμε τη γνωμοδότηση, το Μάρτιο ο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Ίτερ και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια και είναι η πρώτη φορά που ανταλλάσσουμε απόψεις, ε, επιτρέψτε μου στα γρήγορα να σχολιάσω κάποια θέματα σημαντικά. Πιστεύω πως είναι πολύ σχετικά αυτά που είπατε και εσείς κύριε Χατζημαρκάκη και είναι σημαντικό και επιτρεπεί η Ήτρε να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό ε, του τουρισμού. Είναι μια βιομηχανία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 35% της, ε, του ΑΕΠ προέρχεται από εκεί και νομίζω ότι σε αυτή την άποψη πρέπει να το εντάξουμε στις εργασίες μας. 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας με έναν όγκο κύκλο εργασιών που φτάνει το 1, με συγχωρείτε, και με ένα σύνολο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κύκλο που είναι 1,8 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς στην Επιτροπή μας ε, να συμπληρώσουμε κάτι στη γνωμοδότηση. Πολύ σωστά αυτά που είπε ο εισηγητής, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε για κάποιες δράσεις που θα κάνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, δηλαδή βιωσιμότητα και ποιότητα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την κατάρτιση και βέβαια τη σχέση μεταξύ της απέτησης του κλάδου και των κύκλων σπουδών που αυτή τη στιγμή προσφέρονται. Καινοτομία. Καινοτομία και έρευνα, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην ποιότητα και όχι μόνο σε επίπεδο τιμών. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε προωθώντας την έρευνα στην ε, επιστήμη και στις ε, τουριστικές ε, έρευνες για να έχουμε τα αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τον κλάδο και να επιτύχουμε τα αποτελέσματα του κύριου Χατζαμαρκάκη, το οποίο σημαίνει μια καινοτόμα κουλτούρα ε, που θα καλύπτει όλες τις διαστάσεις του τουρισμού. Νομίζω ότι η κοινοτική πολιτική έχει τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να συγκεντρώσει α, τις γνώσεις που έχουμε για τον κλάδο σε ένα σύνολο. Δεύτερον, χρήση της τεχνολογίας για να έχουμε εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να βρουν μια καλύτερη θέση στην αγορά, να γίνουν δηλαδή πιο ανταγωνιστικές. Και τρίτον, να προωθήσουμε τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τουριστικό κλάδο έτσι ώστε η προσφορά να προσαρμοστεί στη ζήτηση στις νέες αυτές συνθήκες. Τώρα για την ε, τεχνολογική πλατφόρμα η οποία θα συγκεντρώνει τα ε, ό,τι γνωρίζουμε για τον κλάδο, αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε εδώ τα όσα θα εντάξουμε, όχι μόνο το που προτείνει η Κομισιόν, αλλά μια πραγματική τεχνολογική πλατφόρμα που θα ε, συγκεντρώνει όλες τις διαστάσεις καινοτομία και της έρευνας. Έχουμε κάποια ακόμα σχόλια που θεωρούμε ότι είναι θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, να δούμε ποιες είναι, τι συνεισφορά μπορεί να έχει ο κλάδος στο να επιτύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ένα θέμα ακόμα, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να πούμε πόσο αναγκαίο είναι να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις που έχουν οι κανόνες που εγκρίνουμε εδώ, ολόκληρο τον τουριστικό κλάδο. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και αργότερα. Θα μπορέσουμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και σε μεγαλύτερο βάθος. Αυτά είναι τα πρώτα που έχω να πω. Και αυτά τα λέω και ως, και ως συγγήτρια εκπροσωπώντας εδώ την πολιτική μου ομάδα. Ευχαριστώ η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την θαυμάσια εισαγωγή σε το σχέδιο της εκθέσεώς του. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με την προώθηση του τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ο τουρισμός ουσιαστικά είναι ένας βασικός οικονομικός παράγων στην Ευρώπη και καλό είναι να σκεφτούμε πως και εμείς θα περιλάβουμε και θα ενισχύσουμε στρατηγικά αυτό το τομέα στο μέλλον. Η δεύτερη παρατήρηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε στο θέμα αυτό και το τρίτο ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η πολιτική γιατί υπάρχουν ε, οι ε, τουριστικές επιχειρήσεις που επιλαμβάνονται και θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτή την προοπτική, να δημιουργήσουμε ε, δραστηριότητες. Οι υποθέσεις, οι επιχειρησιακές είναι θέμα των επιχειρήσεων. Αλλά εδώ συμφωνώ με την κυρία Μαντουρέλ, είναι να υπάρχει ένα έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό στα πλαίσια της αναγνώριση των ε, επαγγελματικών ε, ε, ικανοτήτων και καλό είναι ότι ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, να περιλάβει και τις, ε, τους κανόνες για το ωράριο εργασίας τι γίνεται παραδείγματος χάρη στο room service στον τουρισμό αυτό δεν υπάρχει καθόλου υπάρχουν δηλαδή σε ορισμένους κλάδους ε, οι διάζουσες συνθήκες ε, πρέπει να υπάρχει ε, ίσως ένα συνδυασμός με τις υπηρεσίες υγείας οπότε όμως χρειάζεται κανείς περίθαλψη όλο το 24ωρο και αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη από εργασιακής πλευράς. Επίσης οι Αμερικάνοι έχουν ε, έχουν ε, δημιουργήσει ε, μια φορολογία των τουριστών, tourist και αυτό που με απασχολεί είναι πώς επηρεάζει τους τουρίστες. Υπάρχουν λιγότεροι, λιγότεροι επισκέπτες που θα πάνε στην Αμερική, δεν ξέρω σε τι ύψος είναι, νομίζω 30 δολάρια, αλλά ίσως αν είναι οικογένεια είναι κάτι που θα εξετάσουν. Ε, σε παρακαλώ ε, έλεγξε αν υπάρχουν στοιχεία, αν είχε αρνητική επίπτωση εις την Αμερική, ίσως πρέπει να σκεφτούμε αν και εμείς θέλουμε να το εφαρμόσουμε εις την ε, Ευρώπη. Δεν θέλω υποχρεωτικά να επιβάλλω μια τέτοια φορολογία αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον τουρισμό. Ε, δεν βλέπω άλλους, μάλλον όχι. Τώρα υπάρχει άλλος ένας ομίλητης. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ σύντομα τον συνάδελφο για την παρουσίασή του. με που η Επιτροπή μας ασχολείται με τέτοιο θέμα γιατί μια, εμείς νομίζω ότι ασχολούμαστε κυρίως με τη βιομηχανία. Αλλά δεν πειράζει σε τελική, σε τελική ανάλυση, είναι σημαντικό το θέμα, μας αφορά όλους. Ευχαριστώ και τον ε, προηγούμενο μιλητή, γιατί θέλω και εγώ να μιλήσω για αυτόν τον τουρισμό για λόγους υγείας. Είναι σημαντικό να εναρμονίσουμε τις εσωτερικές σχέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπενθυμίσουμε ότι στο επίπεδο υπηρεσιών προτείνουμε κάτι μοναδικό, δηλαδή τον, του, τουρισμό για λόγους ε, υγείας, ε, τα θερμά λουτρά ε, και τον σχετικό τουρισμό για λόγους θερμών λουτρών. δεν υπάρχουν αλλού α, τέτοιες δυνατότητες. Ε, νομίζω ότι έχει να κάνει με την κουλτούρα μας, με τις χριστιανικές μας ρίζες. Ας τα διαφημίσουμε όλα αυτά, ας διαφημίσουμε και τη δυνατότητα που έχει κάνει να έρθει εδώ για σκι, λόγω του κλίματος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ε, να τα προωθήσουμε όλα αυτά και να εναρμονίσουμε και την ποιότητα των ε, υπηρεσιών. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, θα ήθελα να απαντήσω στην τελευταία πρόταση. Όντως στην Ευρώπη βλέπουμε ότι έχουμε όλο και μεγαλύτερες ασιατικές ομάδες οι οποίες περιδιαβάζουν την Ευρώπη σε 8 μέρες και να αντιμετωπίσουμε την Ευρώπη σαν ένα κοινό τόπο. Για την φορολόγηση υπάρχει τοπική φορολόγηση φορολόγηση, η ε, e αλλά υπάρχουν ε, και άλλες χώρες που έχουν κάποια φορολόγηση όπως η Ισπανία. Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύω ότι είναι πολύ πρόσφατα τα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει ε, φορολόγηση αλλά αυτό που είναι χειρότερο στην Αμερική είναι τα προδιαγραφές ασφαλείας που αποτρέπουν ουσιαστικά τους ε, τουρίστες, πράγμα το οποίο είναι καλό για μας τους Ευρωπαίους, ε, γιατί ε, έρχονται περισσότεροι τουρίστες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα περιλάβω όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν βλέπω κανέναν άλλον, λίγουμε αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας πω ότι τον Ιανουάριο θα δούμε την έκθεση και το Φεβρουάριο θα έχουμε τις τροπολογίες. Έτσι έχουμε φτάσει στο επόμενο θέμα, το οποίο όμως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε, διότι είχαμε προβλέψει την επίσκεψη της Βελγικής Προεδρίας για τις 11.30. Οπότε τώρα θα διακόψω τη συνεδρίαση, ελπίζω όμως ότι δεν θα είμαι μόνος μου σε 11.30 με τη Βελγική Προεδρία. Θα ελπίζω ότι θα χρησιμοποιήσετε το διάλειμμα αυτό για να ξεκουραστείτε σκεφτείτε αλλά μην το σκάσετε. Liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße diejenigen. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και σε, ε, για όσους επανήλθαν ή είναι ακόμη εδώ. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Πολ Μανιέτ, Υπουργό Κλίματος και Ενεργειακής Πολιτικής του Βελγίου. Με συγχωρείτε για τους απόντες. Ε, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα των ε, επιτροπών και γι' αυτό έχουμε πολλές απουσίες. Θα ήθελα όμως να μας ε, δώσετε, να μας την ομιλία σας ώστε όποιος είναι εδώ να μπορέσει να απαντήσει. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ευχαριστώ που είσαστε τόσοι πολλοί για αυτή τη συζήτηση για τον πρώτο απολογισμό της Βελγικής Προεδρίας στα ενεργειακά θέματα. Μου είχατε στείλει στις 12 Ιουλίου ε, να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας. Σήμερα θα σας εξηγήσω Ποιο είναι ο υπολογισμό, ε, προκαταρτικό βέβαια, γιατί το Συμβούλιο Ενέργεια θα γίνει αύριο και κάποια συμπεράσματα και γενικοί προσανατολισμοί θα προκύψουν μόνο μετά το αυριανό Συμβούλιο. Και φυσικά δεν θέλω να προδικάσω τα που θα, τα, όσα θα πούν οι αυριανοί μου αύριο οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω όμω να είμαι πολύ ε, συγκεκριμένο για αυτά που κάναμε και για του προσανατολισμούς στου οποίου έχουμε καταλήξει. Θέλω πριν ξεκινήσω να μιλήσω για τη χρονική στιγμή. Ε, το συζητήσαμε και στις 12 Ιουλίου. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το Συμβούλιο δεν είχε μια μακρά νομοθετική ατζέντα, αλλά ήταν σημαντική η στιγμή της Προεδρίας. Αν δούμε, ε, μέσα σε τι χρονικό ορίζοντα εμείς πήραμε την Προεδρία. Το 2008 ήταν πολύ σημαντική χρονική στιγμή επί Γαλλικής Προεδρίας ε, συμφωνήσαμε για το πακέτο κλίμα και ενέργεια. Μιλάμε για ένα μεγάλο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχεία το 2009 και το 2010 με όλο και μεγαλύτερη ευκρίνεια ε, ξεκίνησαμε προβληματισμό καταρχάς για τον συγκεκριμένο τρόπο που θα υλοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θεσπίσει για το 2020 τι θα κάνουμε, ούτω ώστε να μην μείνουν νούμερα στα χαρτιά, αλλά να γίνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και μέτρα και πώς θα παρατείνουμε τη συζήτηση πέρα από την προοπτική του 2020 για ένα πιο μακροχρόνιο ορίζοντα μέχρι το 2030. Εποφεληθήκαμε από τη σχετική νυνεμία σε νομοθετικό και ρυθμιστικό επίπεδο για να επικεντρωθούμε σε αυτή την ουσιαστική συζήτηση για το ενεργειακό όραμα βραχυπρόθεσμα, μέσα σε 10 χρόνια δηλαδή, και πιο μακροπρόθεσμα, μετά από τη δεκαετία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει ε, στις 4 Φεβρουαρίου μια ειδική σύνοδο που θα την αφιερώσει αποκλειστικά για πρώτη φορά στα ενεργειακά θέματα. Αυτό αποδεικνύει ότι η χρονική στιγμή είναι πολύ σημαντική για το προσδιορισμό του ευρωπαϊκού οράματος. Δεν θα σας απαριθμίσω τις πολυάριθμες συνεδριάσεις που κάναμε και το τι συζητήσαμε, κάναμε δύο συνεδριάσεις υπουργικέ, μία σειρά από συζητήσεις στρατηγικές με εξωτερικούς εταίρους σε ε, Συμβουλίου και ε, μία συνδοκορυφής με τις ΗΠΑ και μία με την ε, Ρωσία στο φόρουμ με τις Επίσης με τους μεγάλους οικονομικούς μας εταίρους, ε, καμία κοσαριά συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας Ενέργειας και πάρα πολλές συνεδριάσεις όπου τέθηκαν πάλι τα θέματα της ενέργειας και όπου ο κόσμος της ενέργειας, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι επιχειρήσεις μας έδωσαν τις απόψεις τους για τα offshore Κάποιε συζητήσεις κάνανε, γυράνε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βιομάζα, ε, πυρηνική ασφάλεια και στι μια μισή, αν δεν έχει τίποτα άλλο να κάνετε, θα γίνει μια σημαντική συζήτηση με του εκπροσώπου της Ευρώπης και του επιστημονικού κόσμου για, την, για το όραμα 2020 στο Παλάτι της Ακαδημίας. Το κάνω λοιπόν έτσι σαν διαφήμιση, ε, γιατί μιλάμε... Γιατί μιλάμε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, περάσαμε τις τέσσερις ε, πρώτες ε, πράξεις ε, εκχώρησης για σημαντικά θέματα της ευρωπαϊκής ιστορίας για τα πλυντήρια, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων και στις 30 Νοεμβρίου δημοσιοποιήθηκαν. Ε, πρόκειται για νέα διαδικασία της Σύνδικης της ε, για τους τομείς αυτούς. Επί της ουσίας τώρα, οι εργασίες μας ε, αφορούσαν τρεις προτεραιότητες ουσιαστικές, την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, τους καταναλωτές και τις επενδύσεις στις υποδομές. Για τους καταναλωτές καταρχήν. Και εγώ και η Βελγική Προεδρία θέλησαν το θέμα των καταναλωτών να μπει στον πυρήνα Τη ε, δουλειά της Βελγικής Προεδρίας της Ένωσης. Εδώ και 10 χρόνια και πάρα από 10 χρόνια ξεκινήσαμε την απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας. Ε, Καιρό είναι να κάνουμε μια πρώτη, ένα πρώτο απολογισμό για να δούμε αν όλε οι υποσχέσει που είχαμε δώσει για τα ωφέλη που θα είχαν οι καταναλωτές, αν σήμερα λοιπόν τι έχουμε υλοποιήσει. Ε, με έκπληξη είδα ότι ο τομέας όπου υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα των καταναλωτών, τελικά είναι το μέσο ενέργειας. Ε, μία σειρά από εργασίε έδειξαν ότι το θέμα της ε, ενεργειακής ανασφάλεια. δηλαδή υπάρχει έντονο, δηλαδή ότι κάποιοι συμπολίτε μας είτε δεν έχουν ε, το ελάχιστο επίπεδο ενέργειας για να ζήσουν αξιοπρεπώς είτε δεν μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμού. Ε, λοιπόν ε, αυτή την ενεργειακή φτώχεια 50 με 125 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Τεράστιο νούμερο αυτή την ε, χρονιά καταπολέμησης της φτώχειας στην Ευρώπη. Επίσης είδα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου προς, με αυτό το θέμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η συζήτηση για τους καταναλωτές θέλουμε να γίνει. Ένας από τους συναδέλφους που έχει την ευτυχία να είναι Μέλο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργεια πάνω από 10 χρόνια, ε, στις 7 Σεπτεμβρίου στο Άτυπο Συμβούλιο είπε ότι πρώτη φορά για 10 μέσα σε δεκα χρόνια που μιλήσαμε για του καταναλωτέ. Για τα πάντα συζητούσε το Συμβούλιο μας, το συμβούλιο μας αλλά ποτέ για καταναλωτέ. Ε, είναι και η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το θέμα των καταναλωτών, γιατί μα το ζητήσατε κι εσεί. Αφιερώσαμε λοιπόν σε αυτό το άτυπο Συμβούλιο ε, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συζητήσουμε και ζητήσαμε από την Κομισιόν ε, να μα υποβάλει μια έκθεση πολύ σύντομα. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή και τι υπηρεσίε τη για να μας εξηγήσει ποια είναι ε, η κατάσταση των καταναλωτών. Το ετοίμασε σε λιγότερο από τρεις μήνες. Ε, δεν θέλω να το απαριθμίσω όλο. Κάποια νούμερα. 13% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, δηλαδή 65 εκατομμύρια Ευρωπαίων, εξοδεύουν δύο φορές περισσότερο για την ενέργεια από το μέσο προϋπολογισμό. Υπάρχει θέμα εδώ διαστρωμάτωσης. 8% των Ευρωπαίων ε, καθιστάνε τις πληρωμές τους για τα, τους λογαριασμούς αυτούς. Ε, υπάρχει ενεργειακή λοιπόν ανασφάλεια. Το Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει συμπεράσματα για το θέμα αυτό. Θα το κάνει αύριο στην άτυπη σύνοδο, ούτω ώστε αυτό το θέμα των καταναλωτών και τη σημασία που πρέπει να δοθεί στους ε, ευπαθείς καταναλωτές να παραμείνει στην ατζέντα. Οι εργασίες θα συνεχιστούν. Καλούμε την Κομισιόν να κάνει τακτικά έκθεση για την ε, εξέλιξη της αγοράς ενέργειας ε, λαμβάνοντα υπόψη την πτυχή των καταναλωτών, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, και θα υποστηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίε, ούτω ώστε να συντονίσουμε καλύτερα αυτό που γίνεται ε, σε επίπεδο απαντήσεων προς του καταναλωτές, δηλαδή το φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια, το φόρουμ του Λονδίνου όπως λέγεται, ή η δικτύωση των Ευρωπαίων διαμεσολαβητών για την ενέργεια, τόσο ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να βελτιώνουν συνέχεια τη λειτουργία της αγοράς. Χαίρομαι που για πρώτη φορά ε, στο έγγραφο στρατηγική για το 2020 που θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο, η Κομισιόν αφιερώνει ένα κεφάλαιο για τους καταναλωτές. Πρώτη φορά γίνεται σε ένα τέτοιο κείμενο. Δείχνει ότι η προσπάθεια αυτή της ε, Προεδρίας να μπει το θέμα των καταναλωτών στην ατζέντα υλοποιήθηκε, ε, τελεσφόρησε. Επίσης, άλλα σημαντικά θέματα, ε, οι επενδύσεις, απαραίτητες επενδύσεις ε, για να έχουμε ευφυείς μετρητές και σε αυτόν τον τομέα ακούμε όλο και περισσότερο αυτά που λέει η Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο. Ε, πριν οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να κάνουμε ε, κοινωνικο-οικονομικές ε, αναλύσεις σοβαρές, ούτως ώστε αυτοί, αυτές οι επενδύσεις να είναι υπέρ και των καταναλωτών, όχι μόνο υπέρ των παραγωγών ας πούμε, αυτών των εφιών μετρητών, παρότι χρειάζεται και αυτό, γιατί πρέπει η εκβιομηχάνηση, η περαιτέρω εκβιομηχάνηση της ε, Ευρώπης να είναι επωφελής και για τους καταναλωτές. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, ένα από τα τρία μεγάλα θέματα του πακέτου ενέργεια-κλίμα, φοβόμαστε ότι η Ευρώπη δεν θα προηγηθεί όπως θα έπρεπε. Ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογική τεχνογνωσία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είμαστε αρκετά μπροστά. Μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ ψηλά επίπεδα ε, και θα ήταν επωφελές όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και των καταναλωτών, ε, θα προωθούσε επίση και τι θέσει απασχόληση και την ε, καινοτομία. Με βάση τι πρώτε εκτιμήσει, όμω δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Μα δείχνει αυτέ οι πρώτε εκτιμήσει ότι αν δεν αλλάξει τίποτα άλλο, αν ακολουθήσουμε τα σημερινά μέτρα, το 2020 η Ευρώπη θα φτάσει σε μία μείωση τη μέση κατανάλωση ενέργεια μόνο κατά 9%. Δηλαδή καθυστέρηση 11% σε σχέση με το στόχο που έχουμε θέσει. Ενώ ορισμένοι εμπειρογνώμονε μα λένε ότι το 2030 με μεγάλη ευκολία μπορούμε, θα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε το 50%. Επομένω πρέπει να κάνουμε ένα Ηράκλειο άλμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μπει πάνω-πάνω στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στο άτυπο συμβούλιο του Σεπτεμβρίου ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και θα είναι το μόνο ε, θέμα επίσης ε, του γεύματο του αυριανού συμβουλίου. Γιατί το, στο γεύμα, όχι γιατί είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά γιατί στο γεύμα ε, συζητάμε πραγματικά ειλικρινά και άμεσα οι διάφορες αντιπροσωπείες. Ε, αυτό το θέμα λοιπόν το βάζουμε στο, στο μεσημεριανό γεύμα για να το συζητήσουμε πραγματικά. Και στις 4 Φεβρουαρίου μαζί με τον Θαρόν τον πρόεδρο και τις υπηρεσίες του, θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου, όπως σας είπα, το Συμβούλιο, ε, η Σύνοδος Κορυφής και θα θέλαμε να μπει ως μέγιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ηγέτη στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Με όλα τα συμπαρομαρτούνται τα θετικά. Ανεξαρτησία, ενεργειακή, ενεργειακός ενεφοδιασμός κτλ. Ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επίσης συμφώνησαν για αυτό το θέμα, για τη συμφωνία ενός ταμείου, το οποίο θα πάρει τα απομεινάρια του σχεδίου ανάκτησης, τα 146 εκατομμύρια τα οποία δεν θα έχουν ε, δαπανηθεί στο σχέδιο ανάκτησης, ε, ανάκαμψης μάλλον, συγγνώμη, που δεν θα έχουν καταναλωθεί ε, από τα κράτη-μέλη για να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές, τις πρωτοβουλίες τους για να προωθήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι ένα ταπεινό βήμα, το αναγνωρίζω, αλλά είναι ένα νέο ταμείο που μπορεί να δημιουργήσει ε, μια, ένα πολύ ενδιαφέρον για την, την εμπλοκή των τοπικών αρχών ε, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί είναι ένα σημαντικό μοχλό αυτέ οι τοπικέ αρχέ. Επίση είναι και πολύ κοντά στου πολίτε και μπορούν αυτέ να, να ευαισθητοποιήσουν πραγματικά του πολίτες για το στόχο αυτό της ενεργειακής αποδοτικότητας. Μεγάλη, τελευταία μεγάλη προτεραιότητα οι επενδύσεις για τις υποδομές. Είναι και ανάγκη για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εφοδιασμού μας σε ενέργεια και ανάγκη για να δημιουργήσουμε μια πραγματική ολοκληρωμένη αγορά και όχι μια, ε, μια συνάθρηση ε, κατακαιρματισμένων αγορών. Ανάγκη επίσης αν θέλουμε να περάσουμε σε αυτή τη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή αλλαγή του ενεργειακού μείγματο, να φτιάξουμε ένα πιο βιώσιμο, πιο αηφόρο ενεργειακό μείγμα, για να εντάξουμε και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για να έχουμε πιο έξυπνα δίκτυα, για να κάνουμε επενδύσει ε, στι υποδομέ. Οι επενδύσει υποδομέ λοιπόν είναι υπό κτονών ουκάνευ. Ε, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα μας λέει ότι θα πρέπει 52 δισεκατομμύρια ευρώ ε, μέχρι το 2020 να δαπανίσουμε κάθε χρόνο αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το 2,5% των ετήσιων δαπανών της Ένωσης και περίπου ε, ισούται με τις επενδύσεις που κάνουμε στις οδικές μεταφορές. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τεράστιες επενδύσεις. Ε, πρόκειται για ένα μαστίγωμα για να προχωρήσουμε. Ήδη είχαμε δώσει 4 ε, δις πιστώσεων, ε, αλλά πολλές από αυτές τις επενδύσεις που είναι στρατηγικής σημασίας για όλους τους λόγους που σας προανέφερα, δεν γίνονται αυθόρμητα στην αγορά, είτε γιατί ε, είναι περίπλοκο το ρυθμιστικό πλαίσιο από χώρα σε χώρα, ε, υπάρχει δυσκολία να βρεθούν χρήματα από τις χρηματαγορές. Θα έπρεπε λοιπόν εμείς να βρούμε αυτό το, αυτούς τους κρίκους που λείπουν, ε, τους τομείς όπου πρέπει να επενδύσουμε και τις τεχνολογίες ε, για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Αύριο η Κομισιόν στο Συμβούλιο ε, θα μιλήσει για τα 59 προγράμματα για τις ε, ε, επενδύσεις ενέργειας και φυσικού αερίου, ύψους 2,365 δις και για το, την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Επίσης, το πάνω από το 96% του ποσού έχει ήδη δεσμευθεί και έχει ξεκινήσει η απορρόφηση. Δεδομένη σημασία του θέματος, ε, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των ε, διαχειριστών των ε, δικτύων ενέργειας και φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, συζητήσαμε με αυτό το θέμα και αύριο το πρωί θα μιλήσουμε ξανά επ' ευκαιρία της ανακοίνωσης της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, κάτι που ενδιαφέρει πολύ τη Βελγική Προεδρία, αύριο, αύριο θα υπογράψουμε στα, στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 10 κρατών, 9 κρατών μελών και ένα τρίτο τρίτου κράτους ε, στη Βόρεια Θάλασσα με σκοπό ε, την ενσωμάτωση της τις ε, εγκαταστάσεις, τις ε, ολικές εγκαταστάσεις offshore. Για να υπάρξει, να προωθηθεί αυτή η πολυεθνική συνεργασία. Το δυναμικό είναι τεράστιο. Ε, μπορούμε μέχρι το 2050 συγγνώμη, να αυξήσουμε κατά 100% το δυναμικό παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει πολύ δυναμικά. Είναι θέματα αυτά τα οποία συζητάμε ε, συνέχεια με την Προεδρία του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε λίγο θα απαντήσω στο σύνολο των ερωτήσεων που θα μου απαντήσετε, αλλά πριν σας δώσω το λόγο θα ήθελα να σας πω ότι χαιρόμαστε που δουλέψαμε πολύ συντονισμένα με την Ισπανική Προεδρία τους που προείδρευσε έξι μήνες πριν από εμά και με την Ουγγρική Προεδρία που θα μας ε, διαδεχθεί την 1η Πρώτου 2011, ο Τόμας Φελέγγι και εγώ ε, και ο Ισπανός ομόλογός μας ε, μέσα στα πλαίσια του τρίου συνεργαστήκαμε καλά για τον προγραμματισμό των Προεδριών. Αύριο το πρωί θα περάσει ουσιαστικά θα δώσουμε, μετά το Συμβούλιο, θα δώσουμε και επίσημα τη σκητάλη στο επόμενο μέλος του τρίου. Αυτά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Υπουργέ, σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσίαση, κατά δεύτερον λόγον για την καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και νομίζω ότι αυτό που είπατε στο τέλος είναι βασικό. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι οι τρεις προεδρίες συνεργάζονται και δεν χρειάζεται κάθε εξάμεινο να ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Οπότε μεταξύ Ισπανίας, εσάς και ελπίζω και της Ουγγαρίας όλα θα, θα πάνε για το καλύτερο ελπίζω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίαση αυτή που μας έκανε. Λάβαμε πάρα πολλές ε, πληροφορίες και για τα όσα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω και να δώσω και ένα κατάλογο θεμάτων που πιστεύω πως θα έπρεπε να συζητήσουμε μελλοντικά ή τουλάχιστον θα έπρεπε να δουν οι Υπουργοί Ενέργειας. Να ξεκινήσω λοιπόν με κάτι το οποίο θεωρώ καθαρά ευρωπαϊκό θέμα. Έχουμε το δεύτερο πακέτο απελευθέρωσης, το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης για την ενέργεια και νομίζω ότι ήδη από το δεύτερο πακέτο και μετά προχωράμε με προβλήματα και δεν ξέρω τι θα γίνει αλλά νομίζω ότι ε, οι υπουργοί θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και θα ήθελα το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα όταν θα συναντηθούν. Νομίζω πως τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον για το θέμα της ενέργειας, έχουμε συζητήσει πάρα πολλά έγγραφα στρατηγικής σημασίας. Θα έλεγα λοιπόν πως δεν θα καταφέρουμε αυτά τα οποία επιδιώκουμε αν παράλληλα δεν τα συνδυάσουμε με κάποιες κατευθύνσεις που θα δώσουμε στη βιομηχανία που θα χρειαστεί να εφαρμόσει τις δικές μας αποφάσεις. Αυτό το οποίο χρειάζομαι λοιπόν είναι να ε, εξασφαλί... αυτό που χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε είναι μια σταθερότητα, ένα πολιτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην έχουμε μεταρρυθμίσεις που θα αλλάζουν το τοπίο κάθε χρόνο. Όταν μιλάμε για στρατηγική του 2020, και μας λέτε τώρα πως έχουμε και μία παράταση για το 2030 αυτής της στρατηγικής. Εγώ θα είμαι πιο φιλόδοξη και θα πω ότι χρειαζόμαστε στρατηγική μέχρι το 2050. Με συνέπεια, με σταθερότητα, ε, τουλάχιστον ε, σε σχέση με τις επενδύσεις. για την χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε σημασία και στο κλίμα και στην αλλαγή του κλίματος. Εσείς είστε υπουργό ενέργεια και κλιματικής αλλαγή. Ε, και γνωρίζετε πως σκοπός μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου αλλά παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την εσωτερική αγορά. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα καθεστώτα στήριξης, μηχανισμούς στήριξης, ε, τους ε, μηχανισμούς ε, προώθησης και όλα αυτά λειτουργούν παράλληλα μεταξύ τους. Πιστεύω πως με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα να σχολιάσετε αυτή μου την παρατήρηση. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως τα διάφορα εργαλεία που έχουμε λειτουργούν με συνεκτικό τρόπο. Για την κλιματική αλλαγή επίσης πρέπει να σας πω πως δεν είμαστε πολύ πετυχημένοι στις προσπάθειες που έχουμε κάνει. Περισσότερες προσπάθειες λοιπόν. Ξέρω πως στο γεύμα με του υπουργού, ξέρω ότι θα σα απαντήσουν. Θα σα απαντήσουν πω ναι, ναι, θα κάνουμε παραπάνω προσπάθειες, ναι, είναι προτεραιότητα, όμω είμαι πεπισμένη πω τελικά δεν θα κάνουν τίποτα. Ρωτώ λοιπόν, έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις με απτά από τους στόχους και αποτελέσματα για να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε πιο, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί ενεργειακά. Υπάρχει κάποιο νομικό δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιβάλλει αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστώ η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είσαστε εδώ σήμερα. και σας ευχαριστώ για όλη την εργασία την οποία έχετε κάνει και ελπίζω θα μπορέσουμε να βασιστούμε και στο μέλλον στην ενεργητικότητά σας προς όφελον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ενέργεια. Χαίρομαι που έχετε αναλάβει το θέμα της ενέργειας και της καταπολέμησης της στόχιας και χαίρομαι διότι θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Επανέρχομαι όμως στο θέμα αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει και στο θέμα των ε, ε, καταναλωτών, δηλαδή την εξοικονόμηση ενεργείας, διότι εχθές έκανε πάρα πολύ κρύο και μπροστά στον Περλεμό είδαμε άνθρωπους οι οποίοι ήταν ντυμένοι σαν πιγκουίνοι. Αυτοί ήθελαν να πούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο φιλόδεξα από πλευράς ενεργείας, από πρωτοβουλίες μέχρι το 2020 και ε, ότι έως τότε οι ε, καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 44 δισεκατομμύρια ευρώ εάν ε, οι καυστήρες μας, ε, εάν τα σπίτια μας ε, ήταν καλύτερα μονομένα, αν οι καυστήρες ήταν πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να γίνουν δηλαδή πολλές προσπάθειες ακόμη και η ενεργειακή πολιτική του Κοινοβουλίου πρέπει να μπορέσει να εφαρμοστεί και να γίνουν ακόμη πολλά που χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει η εξοικονόμηση ενεργείας και μπορούμε να έχουμε εξοικονομήσεις ε, σημαντικές μέχρι το 2020-2030 αλλά τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά ε, ε, δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό πως θα μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε καλύτερο καθεστώς εξοικονόμηση ενεργείας αν δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μέτρα παίρνουμε ένα έτος αναφοράς παίρνουμε το στόχο του 2020 και αν θέλουμε να πετύχουμε πρέπει να κινητοποιήσουμε και να μην αρκεστούμε σε ένα πλαίσιο αλλά σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί επιμελώς. Μιλήσατε επίσης για το Ταμείο. το οποίο θα καταρτιστεί για τις εξοικονομήσεις ενεργείας και πιστεύω ότι αυτή η αποτελεσματικότητα ε, είναι σημαντική και ότι ιδίω μικρά θέματα πρέπει να αναπτυχθούν Εάν προσπαθήσουμε όμως αυτό να προσαρμοστεί στις ανάγκες του καταναλωτή, θα πρέπει ο καταναλωτής όχι μόνο να εξοικονομήσει ενέργεια, αλλά να παράγει επίσης και αυτό είναι πολύ βασικό. Θα ήθελα να ξέρω αν εσείς ενδιαφέρεστε για αυτό το ταμείο, αν πιστεύετε ότι πρέπει να έχει τους αναγκαίους πόρους, να λειτουργήσει σωστά και ε, αν τα θέματα αυτά είναι βασικά για σας, αν μπορεί ε, ε, το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί και αν οι επόμενες προεδρίες θα ακολουθήσουν τα βήματά σας. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την προσοχή ε, με την οποία μας μεταχειρίστηκε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω μέσω ημών ολόκληρη την ε, Βελγική Προεδρία. Νομίζω πως όταν θα αφήσετε αυτά τα καθήκοντα, δεν νομίζω πως θα βαρεθείτε με την διακυβέρνηση του Βελγίου, και σίγουρα θα τα πάνε καλά και οι Ούγγροι, αλλά πραγματικά θα ήθελα να χαιρετήσω τις εξαιρετικές προσπάθειες που κάνετε. Λυπόμαστε λοιπόν, που θα σας χάσουμε λοιπόν για την ε, ενέργεια, την αποδοτικότητα σε ενέργεια. Μιλήσατε για κάποια εργαλεία χρηματοδότησης. Σας παρακαλώ πολύ, ας μην τα ε, πολλαπλασιάζουμε αυτό το τρόπο. Έχουμε παντού υπηρεσίες με διευθυντές, με προέδρους. Είναι δαπανηρά όλα αυτά και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτό το κόστος στον πολίτη μας. Τώρα για την εσωτερική αγορά βασιστήκαμε στους καταναλωτές για να την οικοδομήσουμε και τώρα θέλουμε σε αυτή την εσωτερική αγορά να εντάξουμε και τους παραγωγούς. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των καταναλωτών έτσι ώστε να μην ε, εκπλαγούν οι πολίτες μας από τα αποτελέσματα αυτής της απελευθέρωσης χρειάζεται ενδεχομένως ένα παρατηρητήριο που θα μπορούσε να μας μοιράζει πληροφορίες και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε και κάποια βήματα εμείς στο Κοινοβούλιο με κάποιες προσπάθειες πρωτοβουλίας για την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή στις συγκεκριμένες παραγράφους που αναφέρονται στην ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω πως στηρίζουμε τις δικές σας απόψεις. Και τρίτη παρατήρηση για την ενέργεια και που έχει να κάνει, και έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις που έγινε το 2008 υπό Γαλλική Προεδρία. Ε, για τα θέματα προσπάθειας δέσμευσης του άνθρακα και για τα σύνορα τα οποία προσπαθούσαμε εμείς να θέσουμε ε, στις εκπομπές και τα λοιπά, έχετε εκεί την εντύπωση πως κάτι έχει προχωρήσει και για τις υποδομές δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ανακατευθύσει όλα αυτά. Γιατί βλέπουμε πως υπάρχουν προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προσπαθεί να επενδύσει και δεν θα ήταν καλό να βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την οποία δυσκολευόμαστε να ρυθμίσουμε, μια και είναι και αυτή η χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχει αυτή τη στιγμή ε, rating 3α και νομίζω ότι θα έπρεπε να την αφήσουμε ήσυχη να δραστηριοποιείται ως τράπεζα και όχι ως δικό μας εργαλείο. θα πρέπει οι επενδυτικοί μας δυνατότητες να ενταχθούν ήδη στον προϋπολογισμό για το ΊΤΕΡ και για όλες τις μεγάλες υποδομές και κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες ρώτησα τον Επίτροπο κύριο Ότιγκερ και δεν μου απάντησε τι πιστεύετε, μπορούμε να κάνουμε κοινή αγορά φυσικού αερίου από την Κασπία, δηλαδή να το αγοράζουμε όλοι μαζί. Εσείς σε επίπεδο συμβουλίου συζητήσατε το θέμα αυτό. Και το πιο πολιτικό θέμα στο οποίο πραγματικά δεν λάβαμε απάντηση από τον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ. Εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών είμαστε σίγουροι πως τα ενεργειακά δίκτυα, φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια θα παραμείνουν υπό την κατοχή του δημοσίου. Γιατί βέβαια διαφορετικά δεν θα γνωρίζουμε σε ποιον ανήκουν τα δίκτυα και υπάρχει πρόβλημα πολιτικής δαφάνειας και βεβαίως πολιτικής επιτήρησης. Δεν θέλουμε αύριο να έρθει η Gazprom και να είναι ιδιοκτήτης ε, ε, των δικτύων ή οι Κινέζοι που αγοράζουν τα ελληνικά λιμάνια νομίζω ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους και καλυμμένες ή ακόμα και ανοιχτές επενδύσεις και να έχουμε κατόχους δικτύων ε, που δεν είναι τα κράτη-μέλη. Αυτό θα δημιουργήσει ανησυχία στους πολίτες οι οποίοι πιστεύουν τα δίκτυα αυτά τους ανήκουν. E, Ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Χίμπνερ. Η Προεδρία είναι βαίνει προς το τέλος της. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε και μια σύνοψη των πεπραγμένων. Εσείς πιστεύετε πως ήσασταν επιτυχημένοι στην προεδρία σας. Ποια από αυτά τα οποία παραδίδετε στους Ούγκρους συναδέλφους θεωρείτε ε, πως είναι πρώτης προτεραιότητας. Μιλήσατε για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι. Και είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολλές ανησυχίες. Φαίνεται από τόσα είπατε πως αυτή η οικονόμηση της τάξης του 20% δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέχρι το, 2020 και ε, οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές για 13% των Ευρωπαίων. Λοιπόν, τι δράσεις θα πρέπει να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει πως ο στόχος αυτός της μείωσης του 20% θα έχει θα τον έχουμε πετύχει μέχρι το 2020. Χρειάζεται λοιπόν να εστιάσουμε στις επενδύσεις για να καλύψουμε το περιθώριο απώλειας των δικτύων ή υπάρχουν κάποιες άλλες πηγές ενέργειας στις οποίες θα έπρεπε να στραφούμε. Μήπως χρειαζόμαστε μικρότερες μονάδες οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες πιο κοντά στις καταναλωτές και στις αγορές που εξυπηρετούν. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές στην νομοθεσία μας. Περιμένετε από εμά να αλλάξουμε κάποιους νόμους για να εξασφαλίσουμε πως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, εφαρμοστούν στην πράξη. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουμε είτε στα ψηφίσματά μας είτε στις ε, οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ. Λέω κύριο κύριος Μπαλτσίτης. Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και μας παρουσιάσετε ένα τόσο σαφές όραμα για το τι πρέπει να συμβεί μέχρι το 2050 στον ενεργειακό κλάδο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα έχουμε εξελίξεις και θα τροποποιηθούν και οι θέσεις των οργάνων που εκπροσωπούμε εμείς σήμερα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Οντή. Όταν θα ξεκινήσουν κάποια κράτη-μέλη να απελευθερώνουν τι αγορές τους, αν έχουν ε, μεγάλη συγκαταστάση, για παράδειγμα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας και δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να τα λειτουργήσουν, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ένα στρατηγικός ιδιώτης επενδυτής να ελέγχει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία έχει στήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά ταμεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο εναρμονισμένη πολιτική στο χώρο αυτό. Δεν νομίζετε άλλωστε πω θα έπρεπε ήδη να σκεφτόμαστε ποιε θα είναι οι επιθυμίε και η βούληση των κρατών μελών στο μέλλον έτσι ώστε να συντονιστούμε ευρωπαϊκά. Γιατί νομίζω πως τότε θα ήταν πιο σαφή η κατάσταση. Χθε έκανα την ίδια ερώτηση στον Επίτροπο, κύριο Ότιγκερ, Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα ενεργειακά σχέδια και ενεργικό σχεδιασμό των κρατών μελών μακροπρόθεσμα, να τα κοιτάξουμε σήμερα για να κάνουμε προτάσεις και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, σε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία ενδεχομένως χρειάζονται ε, να βοηθηθούν με κάποιες νέες ιδέες για τη χρήση ανανεώσιμων κτλ. Χρειαζόμαστε χρόνο, χρήμα και στο μέλλον Εάν τα έχουμε αυτά, θα καταφέρουμε να έχουμε μια πιο ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Μπούζεκ, αλλά και το Συμβούλιο, έκαναν κάποιες δηλώσεις για το ότι είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε μια ομάδα δράσης, ένα task force για την αγορά ε, ενεργειακών προϊόντων από τρίτες χώρες. Πιστεύετε ότι θα συσταθεί τέτοια task force και πότε θα αρχίσει να λειτουργεί. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και ε, δίνω τον λόγο στον ομιλητή για να απαντήσει στον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα πάλι να αναφερθώ στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα διότι πολλοί με ρωτάτε από αυτού πράγμα που με χαροποιεί διότι αποδεικνύεται ότι το θέμα αυτό πρέπει να, ε, ε, να σας απασχολεί πολύ ε, και ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο με τις ε, δύο εκθέσεις Φράνσες και ε, Κολάνσα Μπρεζίνκα κινητοποίησε το θέμα αυτό όσον αφορά τους υποχρεωτικούς στόχους αλλά αντί να εντοπιστούμε σε αυτά τα θέματα τα οποία δεν πρέπει να αποφύγουμε δηλαδή τους υποχρεωτικούς στόχους πρέπει να γίνει δουλειά κατά τρόπον ώστε η ενεργειακή αποτελεσματικότητα να, γίνει, να ξαναγίνει αλλά μάλλον να γίνει η πρώτη προτεραιότητα διότι έχουμε ε, ε, εγκαρσίως το διοξίδιο του άνθρακος και καθέτως ε, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα διότι όλοι θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όσο λιγότερο ε, καταναλώνουμε τόσο λιγότερο χρειάζεται να περνά από τους αγωγούς τόσο λιγότερες ανανεώσιμες χρειαζόμαστε δηλαδή κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά από όλε τις απόψεις είναι το πιο χρήσιμο. Κοινό στόχος τον οποίο έχουμε στηρίξει λιγότερο εις το πακέτο και έφτασε η στιγμή να αναθεωρήσουμε. Άρα οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διάσκεψη κορυφής της 4ης Φεβρουαρίου ε, αναφέρεται αυτό το θέμα όπως αναφέρεται ε, και στις προτεραιότητες, στις τρεις-τέσσερις προτεραιότητες αλλά πρέπει να καταστεί πρώτη. Ο στόχος αυτός πρέπει να να διακηρυχθεί από όλα τα θεσμικά όργανα ότι είναι ε, ο στόχος της Ευρώπης να είναι η ηγέτης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας μέχρι το 2020-2030. Μόλις υπάρξουν και άλλοι που συμμερίζονται το στόχο αυτό μπορεί ε, να επεκταθεί σε συγκεκριμένους στόχους που ξεπερνούν τις τωρινές προπτικές. Χρειάζεται βέβαια και ε, μία πολιτική πολιτική τυποποίηση διότι ε, τα πρότυπα έχουν αποδείξει ότι είναι σημαντικά. Βλέπουμε ε, στο αυτοκίνητο παραδείγματο χάρη θεαματικά αποτελέσματα διότι ε, επί χρόνια είχαμε κώδικες καλής συμπεριφοράς που ποτέ δεν απέδωσαν. Μόλις γίναμε πιο πιεστικοί όλα προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει εμείς εμείς ε, στα, στις προδιαγραφές που δεν ήταν δύσκολο να συμφωνηθούν. Οπότε ήταν ένα καλό, ε, μια καλή ένδειξη προς τη βιομηχανία κατά τρόπον ώστε να έχουμε ε, σαφείς ενδείξεις για να ξέρει ο καθένας που πρέπει να επενδύσει και να συνεχίσουμε να τυποποιούμε και να προωθούμε το μίσο που δεν υπάρχουν προδιαγραφές όχι για λόγους γραφειοκρατικούς, όχι για να εναρμονιστεί το σύμπαν, αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε στον τομέα της έρευνας και της βιομηχανίας, πρέπει να γνωρίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε. Έχουμε δημιουργήσει στο Βέλγιο ένα γραφείο περιβάλλοντος και τυποποιήσεως για να δούμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να ξέρουν ότι οι οι βιομηχανίες ε, ε, και οι προσπάθειές τους αναγνωρίζονται και κάνουμε θετικές προσπάθειες στο θέμα της τυποποίησης διότι τώρα οι θερμοσύφωνες, οι καυστήρες τομείς οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί ή στον τομέα της, ε, της ε, ε, οικοδομής και σε ορισμένους κλάδους όπου προβαίνουμε σε σπατάλες ή ανόητες ενέργειες να τυποποιηθεί και να μπορούμε να έχουμε σαφές υποδείξεις ε, ε, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες έχουν πάρα πολλές προδιαγραφές οι οποίες έτσι στηρίζουν και τα ερευνητικά του ιδρύματα και τις βιομηχανίες χωρίς να υπάρχει περαιτέρω νομοθετικό έργο. Μετά η έρευνα και η ανάπτυξη που είναι ένας βασικός τομέας στις ε, ε, έρευνες μας και ε, αυτό είναι ένας τομέας διότι έχουμε καινοτόμες τεχνολογίες αλλά χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες και πρέπει να μπορούν να επεκταθούν εύκολα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία δημοσίων, δημοσίας στήριξης αλλά δεν πρέπει πρώτα να έχουμε τη χρηματοδότηση πρώτα χρειαζόμαστε τους πολιτικούς στόχους, να δώσουμε το σωστό σήμα και μετά να δούμε πόσο θα χρηματοδοτηθούν με βάση τη δεύτερη οδηγία και ε, με την ανάγκη δημοσίας υποχρεώσεως για να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες. Με αυτά τα μέσα δεν θα έχουμε μόνο στόχους αλλά πολιτικούς στόχους για την Ευρώπη. Αν πρέπει να είναι υποχρεωτική ή όχι. Πιστεύω ότι χρειάζεται να είναι υποχρεωτική αλλά δεν έχει λύσει, ε, ε, λήξει η συζήτηση στο Συμβούλιο και έτσι δεν μπορώ εγώ σαν πρόεδρος του Συμβουλίου να σας δώσω μία σαφή δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τα κράτη-μέλη ή τους ενδιαφερομένους, αλλά θέλουμε να έχουμε σωστές εφαρμογές. Και η ερώτησή σας ε, για την εφαρμογή είναι ε, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή ε, το Μάρτιο θα παρουσιαστεί του χρόνου το τρίτο πακέτο. Η Επιτροπή παρακολουθεί την μεταφορά στην Εθνική και την παρακολούθηση και βλέπουμε ότι ε, χωρίς να είναι άκρος υποχρεωτικά είναι χρήσιμο για τα κράτη-μέλη διότι είδαμε ε, προχθές ε, σκεφτήκαμε αν έπρεπε να υποβάλουμε το πρόγραμμα για τις ανανεώσιμες ενέργειες που τελικά υπευλήθη δείξαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο υποχρεωτικός στόχος συζητήσαμε με όλους τους ενδιαφέροντες ενδιαφερόμενους, τις επιχειρήσεις, τους διαχειριστές των δικτύων, τους πολιτικούς. Ε, κινητοποιήσαμε μία δυναμική κοινή ε, περισυλλογής κατά τρόπον ώστε να επιτύχουμε. Και αν όλα αυτά γίνουν και εις ε, την ενεργειακή αποτελεσματική θα μπορέσουν και εντός του τομέα και διαμέσου διαφόρων τομέων αυτό να επιτευχθεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε εάν αυτός ο μοχλός ε, ε, ε, είναι θετικός για να προχωρήσουμε χωρίς να αποτελέσει εμπόδιο για έναν τομέα ή για μια χώρα. Τα κράτη πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν αντί να υπάρχουν ασάφειες και χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι οι χρήσιμοι ακριβείς στόχοι. Μου λέτε συγχρόνως ότι υπάρχουν θέματα που υπερβαίνουν ε, το χρονοδιάγραμμα της Προεδρίας. Δεν θα αποφύγω να απαντήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι όπου δεν έχει ε, αποφανθεί το Συμβούλιο μπορώ να μιλήσω προσωπικά σαν Βέλγιο και όχι σαν Προεδρία της, ε, του Συμβουλίου. Όταν μου ρωτάτε κύριε Οντί για ε, μια φορολογία του διοξιδίου του άνθρακος ε, έχω κάνει το ερώτημα να δούμε αν θα είναι χρήσιμο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν εμπόδια που άπτονται της εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής των κρατών μελών αλλά είδαμε ότι η μεγαλύτερη ελληνική δημιουργήθηκε από το κοινό τιμολόγιο όπου αντισταθμίσαμε ε, το, ε, τη διαφορά μας ε, για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε τα ταμεία συνοχής και τη γεωργική πολιτική. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένας μοχλός προσαρμογής. Αυτό μπορεί να γίνει και για τη φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακος να βοηθήσει τις χώρες που θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη μετάβαση προς τη βιομηχανία για να υπάρξουν μετατροπές σε διαφόρους τομείς για προσαρμογή του κοινωνικού τομέα και ούτω καθεξής. Ε, ίσως ε, ε, μπορεί να αποτελέσει ένα δευτερεύον συγκεκριμένο θέμα αλλά πολύ χρήσιμο στην Ευρώπη πέραν της φορολογήσεως των χρηματαγορών. Και μέχρι σήμερα έχουμε ασχοληθεί με την αλληλεγγύη με τρόπο αμυντικό. Δηλαδή κινητοποιούμαστε ε, για περίπτωση κρίσεως και όλα βαίνουν καλώς. Αξιολογήσαμε με τους ε, ομολόγους Ρώσους στην κοινή διάσκεψη κορυφή ε, που βρισκόμαστε και όλα πάνε καλά. Ξέρω ότι ο κύριος Σέτιγκερ και ο κύριος Ντεγκούχ, το αρμόδιος επίτροπος παρουσιάζουν τις θέσεις μας και χρειαζόμαστε αλληλεγγύη για τα ε, δίκτυα τροφοδοτήσεως Nord Stream, South Stream, Ναμπούκο και ε, τις σχέσεις με τους βασικούς προμηθευτές μας και ε, ομολόγους μας κατά τρόπον ώστε να αποφύγουμε υποδομές που θα υπολειτουργήσουν διότι αν έχουμε υπερβολικούς αγωγούς, ε, θα έχουμε το LNG περισσότερο στις βόρειες ακτές, ε, θα έχουμε κόστη τα οποία θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές και το 230 2040 θα διαπιστώσουμε ότι γίνεται κακή διαχείριση των δημοσίων πόρων. Ε, αντελήφθηκα το μήνυμά σας για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία όμως μέχρι στιγμής επαγρυπνεί και προσέχει πάρα πολύ το θέμα της αποδοτικότητος. Υπάρχει ένας έλεγχος ε, για την τιμολόγηση ε, των ε, τιμών μεταφοράς και έτσι μπορούμε να δούμε πώς θα καλυφθούν αυτές οι επενδύσεις ενώ και εδώ διαβάζω την έκθεση δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι λιγενέση σε όσο αναφορά τις δημόσιες μεταφορές. Μέχρι στιγμής θέλαμε το unbundling, μία, ένα κατακαιρματισμό και από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση. Άρα ε, δεν απαγορεύεται η δημόσια ιδιοκτησία στον χώρο αλλά πρέπει να ελέγχεται. Ας δημιουργήσουμε ανταγωνισμό και αυτό δεν σημαίνει ότι αν είναι ένας ε, χώρος δημόσιος πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο διότι τότε θα ξαναξεκινούσαμε από το μηδέν της συζητήσεις και κύριε Οντή ε, εδώ βρίσκεται η συζήτηση στο επίπεδο του Συμβουλίου και της Επιτροπής και δεν συμφωνούν όλοι. Τώρα, ε, όσον αφορά αν έχουμε πολλά στρατηγικά προγράμματα και λίγες δυνατότητες χρηματοδοτικές δεν νομίζω διότι αν δείτε ε, έχουμε μία λογική χωνιού η οποία είναι σωστή. Καταρχήν είχαμε τους μεγάλους προσανατολισμούς για το κλίμα, την κατάρτιση των στόχων του 2020, πακέτο υποδομών για τις υποδομές, ε, ένα πρόγραμμα για για την επίτευξη των στόχων και μετά δημιουργούμε τις ε, κατάλληλες χρηματοδοτικές δυνατότητες ανά πρόγραμμα. Άρα ε, δεν υπάρχει σύγχυση, έχουμε μία σφαιρική αντιμετώπιση και για μετά το 2020 πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση τώρα για το 2050 για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ε, μία σωστή αντιμετώπιση μακροπρόθεσμα και οδεύοντας προς τα πίσω να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες, την ανάπτυξη και ούτω καθεξής μέσα στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης προοπτικής για να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια εις ε, τις κινήσεις οι οποίες ήδη έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνουν. Και νομίζω ότι έτσι κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις οι οποίες μου είχαν τεθεί. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ εν ονόματι των συναδέλφων για τη συζήτηση, για την ενημέρωση και για την ε, καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμού στους συνεργάτες σας και τις καλύτερες ευχές μου αύριο για τις ε, εργασίες σας. Ευχαριστώ. Οπότε λύεται η συνεδρίαση.